guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie zum öffentlichen. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω στην ε, ακρόασή μας, τη σημερινή. Η εισηγήτρια Ίγκη Εγκλέστερ θα κάνει μια εισαγωγή του θέματος. Καλωσορίζω στην Επιτροπή μας ε, δύο εξαιρετικές προσωπικότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Φερχόγγεν, τον πρεσβύτερο, αντιπρόεδρο επί σειρά ετών και τον νυν αντιπρόεδρο, τον κύριο Σέρκοβιτς. Έχουμε ένα πολύ συναρπαστικό θέμα σήμερα. Το θέμα λοιπόν είναι η αξιοπιστία της εργασίας της ε, Κομισιόν και βεβαίως το θέμα της νέας προσέγγισης ε, της ε, δημόσιας διοίκησης όταν μιλάμε για την Κομισιόν και τις ιδιαίτερες δυσκολίες που σχετίζονται με την περιπλοκότητα ενός συστήματος όπως η Κομισιόν η οποία είναι μάλλον ε, κάτι το μοναδικό παγκοσμίω. Γι' αυτό χαιρόμαστε για το ότι είστε εδώ πέρα. Και βεβαίως ε, το θέμα μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, σε πολλές εκθέσεις, ε, σε στενή συνεργασία με το ελεγκτικό συνέδριο και βεβαίως καλωσορίζω και τους εκπροσώπους του ελεγκτικού συνεδρίου. Το ελεγκτικό συνέδριο επίσης μας έχει ε, πει το πώς μπορούμε να φύγουμε από την ε, διαβεβαίωση αυτή που δίνει σε ε, μια άλλη προσέγγιση η οποία θα βασίζεται στα αποτελέσματα, το λεγόμενο performance-based accounting, ζητήματα δηλαδή που χρειάζονται πολιτική βούληση και βεβαίως δεν εξαρτώνται μόνο από την Επιτροπή μας. Επίσης, οπωσδήποτε σήμερα θα πρέπει να δούμε και το παρελθόν. Γι' αυτό ορίσαμε ως περίοδο την οποία θα δούμε τα 10 χρόνια. Εγώ από το 2009 είμαι εδώ πέρα, παρακολουθώ το τι γίνεται. Αλλά με την ίδια Γκρέσλε, την εισηγητριά μας, ε, ε, η Ίγκερ Γκρέσλε νομίζω πως είναι, ε, μια ειδικός επί του θέματος και θα της δώσω τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε σχεδόν ε, ακριβώς έξι χρόνια πριν η Επιτροπή μας ε, είχε κάνει μια ακρόαση ε, για το ίδιο θέμα. Τότε προσπαθήσαμε να δούμε το τι γινόταν με τη μεταρρύθμιση Κίνοκ που ακολούθησε την παρέτηση της Επιτροπής Σαντέρ. Τέσσερα θέματα έχουμε. Δεν θα τα πω με τη σειρά βεβαίως ε, που είναι στην ημερησία διάταξη. Το θέμα είναι τι κάνουμε με την αποκέντρωση και την εξωτερική ανάθεση αρμοδιοτήτων από όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 48 υπηρεσίες και γενικές διευθύνσεις με δικό του site, ε, ε, δική τους διεύθυνση προσωπικού, επικοινωνίας, προϋπολογισμού και βεβαίως υπάρχουν 37 εξωτερικές υπηρεσίες, 7 κοινοπραξίες και 6 εκτελεστικές υπηρεσίες ε, που απασχολούν 1625 υπαλλήλους. Το 2007 είχαμε μόνο 4 εκτελεστικές υπηρεσίες και 582 υπαλλήλους. Οπότε το θέμα της ε, γραφειοκρατίας δεν είναι μόνο ζήτημα ε, αρμοδιοτήτων οι οποίες αλληλεπικαλύπτονται. Υπάρχει λοιπόν ένα πάρα πολύ σημαντικό έγγραφο που μας βοηθήσει, θα μας βοηθήσει εδώ πέρα, είναι το, οι εκθέσεις ε, staff screening όπως λέγονται, οι οποίες εκδίδονται κάθε 30 Απριλίου. Είναι πάρα πολύ σημαντική αλλά δυσανάγνωστη πηγή ε, των αποτελεσμάτων. Ποια είναι τα αποτελέσματα λοιπόν το 2007 32% των ε, υπαλλήλων της Κομισιόν είναι, εργάζονται σε μια διοικητική ή υποστηρικτική εργασία. Και το δύο, τα δύο τρίτα από αυτούς ε, είναι στις ε, κεντρικές ε, γενικές διευθύνσεις, δηλαδή προσωπικού και επικοινωνίες. Και βεβαίως ε, εγώ είχα κάποιες διαφωνίες με τις κομισιόν το πώς τα υπολογίζουν αυτά. Εγώ λυπούμαι για το ότι αλλάζουν συνεχώς οι κατηγορίες, κατά το οποίο κύριε Σεύκοβιτς οδηγεί στο ότι δεν υπάρχει ακριβώ η διαφάνεια την οποία θα θέλαμε υπήρχε η προσπάθεια να αλλάξει η σχέση μεταξύ κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών. Τι ρόλο παίζει η Γενική Γραμματεία, τι ρόλο πρέπει να παίζει. Να δεν λέει η εκπρόσωπη μας πως ε, η Γενική Γραμματεία πηγαίνει να γίνει ένα γραφείο του Προέδρου και αυτά είναι οι ζητήματα στα οποία θα ήθελα να απαντήσει ο κύριος ε, Σεύκοβιτς. Επίσης, το δεύτερο ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή πώς η Επιτροπή, δηλαδή το πολιτικό πλέον επίπεδο, ε, λαμβάνουν ε, αποφάσεις προϋπολογισμού και λογοδοτούν. θεωρητικά βεβαίως ε, αυτά γιατί στην πραγματικότητα δεν υπογράφει και δεν είναι υπεύθυνος για τον προϋπολογισμό ο Επίτροπος αλλά ο Γενικός Διευθυντής του. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω τι γίνεται με αυτό. Από ό,τι φαίνεται, ε, αυτός ο οποίος μας δίνει λόγο κάθε έτος είναι ο Γενικός Διευθυντής με την ετήσια έκθεση και βεβαίως ε, μας λέει ότι ενημέρωσε τον Επίτροπο. το θέμα είναι τι αλλάζει με αυτή την ε, κατάσταση. Δηλαδή, τι γίνεται στην πράξη. Το ΩΣΔΕ το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου επί μία δεκαετία δεν λειτουργούσε στην Ελλάδα. Μετά ανακαλύπτουμε πως δεν λειτουργεί από το 2008 στη Βουλγαρία και από το 2010 δεν λειτουργεί στην Πορτογαλία. Το πρόγραμμα της αλληλείας έχει προβλήματα στη Γερμανία από το 2010 και τα διαρθρωτικά ταμεία βεβαίως ξέρετε πως ε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι προβληματικά στην Ισπανία και την Ιταλία. Οπότε τι σημαίνει τελικά αυτή η ευθύνη ή τι αλλάζει στην πράξη. Και κατά πόσο μπορούν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση οι επίτροποι κανονικά. Αυτός ο οποίος έχει την εξουσία είναι αυτός ο οποίος ε, δίνει τα λεφτά. Οπότε φαίνεται αυτοί οι οποίοι κέρδισαν από τη μεταρρύθμιση Κίνοκ ήταν οι γενικοί διευθυντές. Κάτι θα μπορέσει να μας είχε ο Φερχόγγεν ο οποίος ήταν ο μόνος ο οποίος έκανε θέμα αυτή ακριβώς την τεταμένη σχέση μεταξύ γενικών διευθυντών και πολιτικής ηγεσία. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που ξανά ήρθατε, ε, κύριε Επίτροπε, για να μας μιλήσετε για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο το ξέρετε από μέσα. Εδώ πέρα τώρα δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε κάποιον, απλά θέλουμε να δούμε πώς ε, λειτουργούμε ως διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα ανησυχώ για το ότι στα βασικά και εδώ πέρα φτάνουμε στο τρίτο θέμα στα βασικά λοιπόν της διοίκησης υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο διορθώσεων. Γιατί δεν υπάρχει ένα ενιαίο διοικητικό δίκαιο εντός της, ε, εντός της διοίκησης το οποίο θα ισχύει και για την Κομισιόν και για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Και βεβαίω υπάρχει και διαφορετική ερμηνεία. Όμως θα πρέπει η διοίκηση να προσφέρει μια ασφάλεια δικαίου και βεβαίω να είναι προβλέψιμη στην δραστηριότητά της. Γι' αυτό θα ήθελα να σα παρακαλέσω κύριε Σεύκοβιτ, για λόγους αξιοπρεπίας, ε, αξιοπρέπειας της ε, Κομισιόν να βάλετε αυτό το ζήτημα στην... Ε, στον ε, κατάλογο των ε, προσεχών προτεραιοτήτων της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως έχω περάσει πάρα πολύ χρόνο ακούγοντας τα παράπονα των επιχειρήσεων που δεν έχουν καμία δυνατότητα όταν έχουν διαφορετική και αιτιολογημένη νομικά άποψη να μπορέσουν να την υποστηρίξουν ενώπιον των αποκεντρημένων υπηρεσιών. Και κάτι τελευταίο, αλλά ουσιαστικό. Μια δημοκρατική Ευρώπη επίσης χρειάζεται μια κοινοβουλευτική βάση για το τι γίνεται σε σχέση με τους επιτρόπους. Δεν υπάρχει ένα, μια νομοθεσία η οποία θα ήταν ανάλογη με την νομοθεσία περί ευθύνης υπουργών που έχουμε ε, στο εθνικό επίπεδο. Και επίσης ε, οι αμοιβέ των ε, επιτρόπων ορίζονται σε έναν κανονισμό του Συμβουλίου από το 1967 με βεβαίως τελευταία αλλαγή το 2012. Θεωρώ επίσης πως ε, ένα άμεσα ερετό κοινοβούλιο μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα στον ε, τομέα αυτόν. Επίσης χαίρομαι για το ότι εκπροσωπείται και ο κύριος ε, Σεμπαστιάνη εδώ πέρα και θα ήθελα να χαιρετήσω και τον καθηγητή, τον κύριο Χουσέιν ε, Κασίν και τον καθηγητή Μιχαήλ Μπάουερ, ο οποίος βεβαίως ε, δυστυχώς δεν είναι εδώ πέρα σήμερα και εκπροσωπείται από τον κύριο Στέφαν Μπέκερ. Μην ξεχνάμε πως είχαμε τις ακροάσεις του 2007 οι οποίες ξεκίνησαν την μεγαλύτερη μελέτη που είχε υπάρξει ποτέ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε το θέμα είναι ακριβώς που λαμβάνονται οι αποφάσεις και ποιο ρόλο παίζει η Γενική Γραμματεία σε όλο αυτό τον σχηματισμό αυτόνομων κέντρων λήψης αποφάσεων η κυρία, η δόκτωρ Άνριχτ Βίλε του Πανεπιστημίου του Λάιντεν επίσης έχει συνεισφέρει πάρα πολλά σε αυτόν τον τομέα. Σας ευχαριστώ. Πριν περάσουμε στους ε, υπόλοιπους ομιλητές. Θέλω να πω πως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον εμείς που λαμβάνουμε τις αποφάσεις να διαβάζουμε καμιά φορά και ε, επιστημονικές ε, μελέτες, αν και βεβαίως από ό,τι φαίνεται συχνά κινούμαστε με βάση την αρχή της απροσδιοριστίας του Χάιζενμπεργκ. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Επίτροπο, ο οποίος θα παρέμβει με τίτλο «Ποιος έχει τον τελικό λόγο, ο Επίτροπος ή η διοίκηση» Ο κύριος Φερχόγγιν. σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι ξανά εδώ πέρα. Ε, πραγματικά ε, επί μια δεκαετία είχα απολαύσει την συνεργασία με το Κοινοβουλίο, κατά οποίο δεν μπορώ να πω για όλα τα θεσμικά όργανα. Και ε, αναρωτήθηκα γιατί καλέσατε εμένα. Τελικά ήταν α, σαφές, έγινε σαφές χτες. Το θέμα λοιπόν είναι πώς θα διασφαλίσουμε το ότι η πολιτική θα έχει τον πρώτο λόγο γιατί ο γραφειοκρατικός μηχανισμός γίνεται όλο και μεγαλύτερος και από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια προσπάθεια να κατευθύνει την πολιτική ηγεσία. Κοιτάξτε, Εγώ δεν ε, κατέληξα σε αυτό το θέμα αναζητώντας ένα ζήτημα ε, για να ασχοληθώ. Απλά η πολιτική μου ε, σταδιοδρομία είχε ξεκινήσει με μια επιταετή θητεία σε μια θέση και ήταν η πιο σημαντική. Θα έλεγα ότι είχα ασκήσει περισσότερη επιτροπή όχι ως επίτροπος, όχι ως υπουργός. Τη μεγαλύτερη εξουσία την είχα α, 7 ε, χρόνια ως υπάλληλο όπου ενημέρωνα τον Υπουργό, έκανα προτάσεις, ε, του έλεγα τι να κάνει, του έλεγα ποια είναι τα θέματα που έπρεπε να τον απασχολήσουν χωρίς να έχω εγώ προσωπική ευθύνη για το αποτέλεσμα αυτών των πράξεων. Και από τότε με απασχολεί αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα λοιπόν του πολιτικού ελέγχου επί της διοίκησης δεν είναι ιδιαίτερο και μοναδικό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει παντού. Και παρόλα αυτά πρέπει να δούμε τις ιδιαίτερες πτυχές της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής γιατί είναι ιδιαίτερη για ιστορικούς λόγους και για θεσμικούς λόγους και δημιουργεί κάποια θεσμικά προβλήματα που δεν υπάρχουν αλλού. Το ζήτημα λοιπόν είναι πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε κάποιες διαδικασίες με τις οποίες θα επιβάλλεται στην καθημερινή ε, εργασία των υπηρεσιών η πολιτική βούληση Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Κομισιών. Απλές συμβουλές και συνταγές δεν έχω γιατί βεβαίως η αλληλεπίδραση αυτή δεν ε, ακολουθεί την ε, λεγόμενη αρχή Yes Minister Θα θυμάστε βεβαίως την γνωστή σειρά όπου ήταν μαριονέτα στα χέρια των υπαλλήλων η πολιτική. Μπορεί να είναι διασκεδαστικό αλλά δεν ε, περιγράφει την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να αναφερθώ σε, στους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ταυτόχρονα έχει μία συνέχεια και μία ασυνέχεια. Πρώτα απ' όλα ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια η Κομισιόν. Δεν υπάρχει ένα σώμα της Επιτροπής το οποίο αναλαμβάνει εξουσία με κάποιες προγραμματικές δηλώσεις όπως γίνεται στο εθνικό επίπεδο η Κομισιόν λειτουργεί με βάση το εκτεταμένο βεβαίως ευρωπαϊκό δίκαιο. Προκύπτουν λοιπόν νομοθετικές προτάσεις που έχει επεξεργαστεί και η προηγούμενη Επιτροπή. Ο προϋπολογισμός επίσης έχει προκαθοριστεί μέσω των 7 ετών προγραμμάτων και υπάρχουν και προσδοκίες και μακροχρόνιες συζητήσεις είτε στο Κοινοβούλιο, είτε στα κράτη-μέλη, είτε με τους λεγόμενους ε, ενδιαφερόμενο. Καμία κομισιόν λοιπόν δεν ξεκινάει σε κενό. Κανένα μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορεί να τα ξέρει όλα αυτά. Δεν είναι σε θέση, ανεξαρτήτως του ποια πολιτική σταδιοδρομία είχε. Και βεβαίω δεν μπορεί να τα ξέρει όταν προετοιμάζεται για την ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ακρόαση αυτή, όπως ε, ξέρετε, είναι αποφασιστική σημασίας, καθώς μπορεί κάποιος να αποτύχει σε αυτήν. Τι έκανα εγώ, λοιπόν. Πρέπει να βασιστεί ο Επίτροπος στη Συμβουλή, στην γνώση, στην εμπειρία, θα έλεγα στη συλλογική μνήμη των υπηρεσιών της Κομισιόν, οι οποίοι ξέρουν το σχετικό δίκαιο, δεν έχουν μια στενή εθνική σκοπιά και γνωρίζουν και τις προσδοκίες του Κοινοβουλίου και της ευρωπαϊκής ε, κοινή γνώμης. Και βεβαίω υπάρχει μια πάρα πολύ, αρχική, ε, πολύ εντατική αρχική φάση εργασίας με τον ε, νέο επίτροπο. Αλλά βεβαίως εκεί πέρα ακριβώς παρατηρούν οι υπάλληλοι το προσωπικό, το εάν ο νέος επίτροπος πραγματικά ενδιαφέρεται για τα θέματα, αν έχει την πνευματική ικανότητα να παρακολουθήσει δύσκολα ζητήματα, εάν θέτει τις σωστές ερωτήσεις, εάν είναι ικανός για ομαδική εργασία κτλ. κτλ. Η δική μου εμπειρία στον τομέα αυτών είναι πολύ θετική. Εγώ θεωρώ πως μου έδωσαν καλές συμβουλές, αλλά είχα και την ε, ελευθερία να κάνω αυτό το οποίο θέλω. βεβαίω, βεβαίως χρειάζονται πάρα πολλά ε, πράγματα για να ε, σχηματιστεί μια πραγματική ομάδα. Ανεξαρτήτως των εμπειριών που έχει κανείς, διαπιστώνει γρήγορα πως η δουλειά του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου δεν συγκρίνεται με ένα Υπουργείο. Κυρίως γιατί η Κομισιόν λειτουργεί ως συλλογικό όργανο και άρα χρειάζεται τη στήριξη της πλειοψηφίας και κυρίως ε, του Προέδρου για να μπορέσει να κινηθεί ένας επίτροπος. Επίσης είχαμε ακριβώς ε, τα τελευταία χρόνια έναν συγκεντρωτισμό την, ε, της λειτουργίας κομισιών ή όπως λέγεται αυτό το upstream coordination. Αυτό βέβαια σχετίζεται με το μέγεθος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά Δεν ξέρω αν είναι θετικό, γιατί περιορίζεται πάρα πολύ, όπως είπα, ο συλλογικός χαρακτήρας της ε, Κομισιόν. Αλλά εξακολουθεί, όπως είπα, να δράω ένα σώμα ε, το σύνολο των επιτρόπων. Επίσης, ο Επίτροπος πρέπει να εκπροσωπεί και τα συμφέροντα των κρατών μελών και, και <coughs> ε, του Κοινοβουλίου. Βεβαίω, στο Κοινοβούλιο τα πράγματα είναι διαφορετικά από τα εθνικά κοινοβουλία γιατί δεν υπάρχει συμπολίτευση, δεν υπάρχει θα λέγαμε μια κυβερνητική πλειοψηφία αλλά η πλειοψηφία είναι κάτι το οποίο αναζητάμε κάθε φορά κατά περίπτωση. Οπότε εδώ πέρα το ζήτημα γίνεται πολύ πολύπλοκο γιατί ο καθένας έχει βεβαίως και την ιστορία του, τη γλώσσα του, την προσωπικότητά του κτλ. Όταν ήμουν λοιπόν αντιπρόεδρος ε, και αρμόδιος για την ε, βιομηχανία ζήτησα να μου κάνουν όλες τις προτάσεις στα αγγλικά. Ο δε επίτροπος ο οποίος με διαδέχτηκε ε, ζήτησε ενημέρωση στα γαλλικά. Βεβαίως Εντάξει, αυτά σιωπηλά τα βλέπουν οι υπηρεσίες, αλλά αντιλαμβάνονται αν κάποιος δουλεύει σκληρά, εάν μπορεί να αντιληφθεί τα ζητήματα, εάν διαβάζει καν τους φακέλους που του στέλνουν, κάτι το οποίο ε, δεν συμβαίνει κατά κανόνα από τη δικιά μου πείρα και βεβαίως παρατηρούν το εάν έχουν να κάνουν με κάποιον ο οποίος έχει το θάρρος της γνώμης του ή ε, με κάποιον ο οποίος προτιμάει μια άνετη ζωή και κάνει ό,τι του λένε. Είμαι λοιπόν πεπισμένος πως οι υπηρεσίες προτιμάνε ένα επίτροπο ο οποίος εργάζεται σκληρά. Είμαι επίσης πεπισμένος πως χρειάζονται κάποια αντίδραση και καλύτερο είναι εξ αρχής να διαμορφώνεται συλλογικά η πολιτική για να γνωρίζουν όλοι ποιοι είναι οι στόχοι και να μπορούν να είναι στήριξη για τη στήριξη του Επιτρόπου. Αλλά επίσης έμαθα πως αυτό δεν ισχύει βεβαίως και για όλο το προσωπικό. Αναγκάστηκα να διώξω έναν υπάλληλο ο οποίος αγνοούσε τελείως ε, τις ε, επιθυσμίες μου και θεωρούσε ότι ήταν πάνω από όλους. Είχα προτείνει τότε τη διαδικασία του άρθρου 50 και ε, αρχικά μετατέθηκε, αλλά και στη νέα του γενική διεύθυνση ο άνθρωπος αυτός ε, είχε την ίδια συμπεριφορά. Τελικά όμως απολύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως αυτή αυτό ήταν ε, ένα ακραίο παράδειγμα. Εντάξει, πρέπει να το πω αυτό. Δεν. Ε, επίσης δεν μπορώ να ισχυριστώ πως όλοι οι υπάλληλοι ήταν πάντα ικανοποιημένοι από τις αποφάσεις μου, αλλά ακολουθούσαν πιστά και με τρόπο δίκαιο αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουν. Το πραγματικό πρόβλημα θεωρώ ήταν πως ε, οι πάλι δεν αναγνώριζαν ένα πολιτικό πρόβλημα ως πολιτικό. Δηλαδή ζούσα συνεχώς το ίδιο και το ίδιο πράγμα. Δεν είχαν συχνά αντίληψη της έκτασης των προβλημάτων. Πράγματα πήγαιναν στραβά επί σειρά ετών, χωρίς κανείς να τα διορθώνει. Και αυτό συμβαίνει συχνά γιατί δεν αντιλαμβάνονται ένα πρόβλημα ως πολιτικό οι υπηρεσίες. Και δεν του περνάει καν από το μυαλό ε, ότι θα μπορούσα να ενημερώσω το γραφείο του Επιτρόπου. Και είχα πολλές περιπτώσεις όπου επί σειρά ετών δεν λαμβάνονταν αποφάσεις ή γίνονταν ανεκτές ε, λανθασμένε ε, καταστάσεις γιατί κάποιος είχε λάβει την απόφαση πως αυτό το ζήτημα δεν είναι πολιτικό, δεν έχει πολιτική σημασία. Και αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να λυθεί με την δομή της ε, Κομισιόν. Δεν είναι δυνατόν επίσης να γίνει το, το γραφείο του Επιτρόπου τόσο μεγάλο ώστε κάθε μονάδα να ελέγχεται από το γραφείο αυτό. Και δεν το θέλουμε κιόλας έτσι. Αλλά ακριβώς εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πως τα πολιτικά ζητήματα δεν αναγνωρίζονται ως τέτοια. Έτσι, δεν είναι θέμα κακής βούλησης. Δεν θέλει κανείς να, να βλάψει τον Επίτροπο, απλά σκέφτεται ο κόσμος ότι αυτό είναι δική μας υπόθεση, θα το λύσουμε. Και υπήρχαν προβλήματα που θα μπορούσαν να λυθούν ε, με ένα απλό τηλεφώνημα, έτσι, με, σε έναν υπουργό ή σε έναν άλλον επίτροπο. Και ε, χρόνιζαν αλλά αυτό δείχνει ακριβώς την σημασία του να αναγνωρίζουν οι πολιτικοί διευθυντές το τι είναι πολιτικό πρόβλημα και τι όχι. Και βεβαίως αποστολή του Επιτρόπου είναι να ξεκαθαρίσει το τι θεωρεί ο ίδιος πολιτικό ζήτημα. Με βάση λοιπόν την εμπειρία μου μπορώ να πω πως Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω στενής ε, συνεργασίας και επαφής ε, του Επιτρόπου και των υπαλλήλων στη Γενική Διεύθυνση. Είχα ακούσει πως ε, προ της Επιτροπής Πρόντι δεν ήταν σύνηθες να συναντάει ο Επίτροπος το Γενικό Διευθυντή. Και υπήρχαν ε, οι απολύτως απαραίτητες ε, συναντήσεις ε, με τον Γενικό Διευθυντή και τους Διευθυντές. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια δική της κουλτούρα λειτουργίας. κατά κανόνα προσλαμβάνει νέους ταλαντούχους ανθρώπους, οι οποίοι βεβαίως έχουν ως ε, πραγματικότητα και περιβαλλούν ακριβώς την ε, Κομισιόν. Τα πράγματα και η κατάσταση στη χώρα τους είναι συνήθως διαφορετική και βεβαίως διαφέρουν και ε, οι κοινωνικές καταβολές κτλ. Αλλά οι επίτροποι στην αρχή δεν παίζουν κανένα ρόλο για αυτούς τους ανθρώπους. Περισσότερη σημασία έχει ο τιματάρχης τους και οπωσδήποτε μετά ο διευθυντής τους. Ταυτόχρονα πολλοί νέοι άνθρωποι αναλαμβάνουν πολύ δύσκολους ε, φακέλους, ε, τους οποίους, ε, συνε... τους οποίους συζητούν με εκπροσώπους των κρατών μελών, των κοινοβουλίων κτλ. Δηλαδή έχουν πάρα πολύ συχνά τεράστιες ευθύνες εξ ονόματος της Κομισιόν. Και ακούμε συνέχεια, η Κομισιόν έκανε αυτό, η Κομισιόν έκανε εκείνο. Η Επιτροπή όμω, δηλαδή η Επίτροπη, το Σώμα των Επιτρόπων, δεν μπορεί να μην έχουν ασχοληθεί ποτέ με ένα ζήτημα. Έτσι. Και βεβαίω ο καθένα από αυτού θέλει να κάνει μια σταδιοδρομία. Και βεβαίω ε, σταδιοδρομία δεν γίνεται μέσω του πολιτικού προϊσταμένου, αλλά μέσω τη φυσική ηγεσία, ε, θα λέγαμε. Γιατί από ένα επίπεδο και πάνω φτάνει κανείς να έχει επαφές με τον Επίτροπο. Και βεβαίως εκεί πέρα αρχίσουν να αναπτύσσονται διάφορες σχέσεις και η δικτύωση είναι το α και το ω της Κομισιόν. Όποιος είναι καλός στην δικτύωση μπορεί να διεκπεραιώσει πράγματα επιτυχώς. Βεβαίως τέτοιους ανθρώπους τους χρειάζεται ο κάθε επίτροπος, αλλά η δικτύωση αυτή, ξέρετε, δεν απέχει πάρα πολύ από τα κολλητηλίκια, θα λέγαμε, και κάποια στιγμή θα μπορούσε να φτάσει κάποιος να δώσει προτεραιότητα σε, ε, αυτό, σε αυτή την πτυχή. Και οπωσδήποτε ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ε, κάποια στιγμή ο Επίτροπος θα φύγει και ο κάθε υπάλληλο θα μείνει με τους συναδέλφους του. Και πρέπει να το λαμβάνει και αυτό υπόψη. Και μην ξεχνάμε, δηλαδή αυτό μπορεί να οδηγήσει πως στο ότι αν κάποιος ήταν, ε, είχε εργαστεί για ένα αφεντικό το οποίο τελικά ήταν μη δημοφιλές μπορεί να τιμωρηθεί και να καταλήξει σε μια τελείως αδιάφορη δουλειά. Οπότε, να σας πω, εγώ το 1999 λίγες εβδομάδες μόλις είχα αναλάβει ε, καθήκοντα και ο Γενικός μου Διευθυντής έδωσε μια συνέντευξη σε ένα ευρωπαϊκό μέσο ενημέρωσης και είπε κάτι το, το τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο θεωρούσα εγώ. Και τι έλεγε, έλεγε, πολιτική χαράζουμε εμείς, οι γενικοί διευθυντές. Ο Επίτροπος είναι για να τα παρουσιάζει, να τα εξηγεί. Ναι, ναι, αυτό είχε πει. Και βεβαίω αυτό οδήγησε ε, σε μια πάρα πολύ έντονη συζήτηση με τον Γενικό Διευθυντή και τελικά είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Αλλά τελικά δεν το είχε ε, αποδεχτεί ποτέ. Και αν μου πείτε, ε, αν μου πείτε από πού προέρχεται αυτό, εγώ θεωρώ πως προέρχεται από τον καιρό του Ζακ Ντελόρ. Είναι μια νοοτροπία της εποχής Ντελόρ ειδικά σε πολύ υψηλό βαθμό υπαλλήλους, οι οποίοι είναι πεπισμένοι πως αυτοί είναι οι μόνοι οι οποίοι, είναι, ε, οι οποίοι αντιλαμβάνονται μακροπρόθεσμα το ευρωπαϊκό κοινό καλό. Και ε, έβλεπα πως ε, συχνά οι γενικοί, διεθ, οι γενικοί διευθυντές αντί για το εμείς ήταν ε, στο εγώ. Βεβαίως εντάξει έχουν πάρα πολύ δύσκολη υπεύθυνη δουλειά, έχουν την ευθύνη για μια ολόκληρη γενική διεύθυνση, έχουν την πλήρη ευθύνη για τον ε, προϋπολογισμό, έχουν τους πολιτικούς που αλλάζουν συνέχεια και συχνά είναι οι άνθρωποι κλειδιά, οι συνομιλητές για τρίτους. Γιατί μην το ξεχνάμε, για τον έξω κόσμο για ανθρώπους οι οποίοι συναλλάσσονται με την Κομισιόν, ο Γενικός Διευθυντής είναι ο σημαντικότερος εκπρόσωπος. Και εκπροσωπεί βεβαίως και τη συνέχεια της υπηρεσίας και πάρα πολλοί θεωρούν τον Γενικό Διευθυντή ή τη Γενική Διευθύντρια ε, σημαντικότερο από τους επιτρόπους. Εγώ θεωρώ πως το γερμανικό μοντέλο της πολιτικής διεύθυνσης ε, θα ήταν καλύτερο. Και μάλιστα θεωρώ πως θα ήταν καλύτερο οι επίτροποι να έχουν περισσότερες δυνατότητες ε, πολιτικής εκπροσώπησης. Όπως πρότεινε παραδείγματος χάρη η Επιτροπή Εξωτερικών για τον τομέα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω κάτι άλλο. Πρέπει να αντιληφθούμε επίσης πως οι υπηρεσίες κομισιών έχουν ε, ελάχιστα ερεθίσματα από έξω. Οι εθνικοί υπάλληλοι είναι αποσπασμένοι για λίγο χρόνο και με την εξαίρεση βεβαίως ε, τα γραφεία των επιτρόπων δεν είναι ποτέ σε θέσεις ε, κλειδιά. Και βέβαια ε, αυτό είναι ζήτημα όταν μιλάμε για ανάγκες και κοινωνικά προβλήματα στα κράτη-μέλη. Και συχνά παρατηρεί αργά η Κομισιόν ε, το ε, το κοινωνικό τίμημα της διαχείρισης της κρίσης του χρέους. και εγώ θεωρώ πως ε, και το είχα, στείλει μάλιστα ανθρώπους να δουλέψουν ε, σε επιχειρήσεις, να κάνουν μαθητεία σε επιχειρήσεις για να δουν τους ανθρώπους οποίους εξυπηρετούν. Έπρεπε να δείτε το, τη φάτσα ενός υπαλλήλου, τον οποίον έστειλα να δουλέψει σε φούρνο και ξύπνα για 3 ώρα το πρωί. Εξακολουθούν βεβαίως ε, εντός κομισιών πάντα να θεωρούν πως η περισσότερη ολοκλήρωση θα έρθει με όλο και περισσότερους ε, κανόνες. Πραγματικά ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να παλέψω. Βεβαίως Σήμερα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχει και η πρωτοβουλία της λεγόμενης καλύτερης νομοθεσίας και μιλάμε βεβαίως εντωμεταξύ για smart regulation, αλλά εντωμεταξύ έχει πέσει πάρα πολύ ο ρυθμός. Οπότε το ζήτημα της δεν είναι απλά να υπάρχουν κανόνες, αλλά ενιαίοι e κανόνες για όλους. Ε, και υπάρχουν πολλά παραδείγματα που δείχνουν πως είναι αναγκαίο να υπάρξει μια νέα σκέψη στην ε, καθημερινή εργασιακή ζωή ε, για να περάσει η αντίληψη πως καμιά φορά η ευελιξία είναι καλύτερη από την ε, εναρμόνιση, ειδικά παραδείγματο χάρη στον τομέα τη εσωτερική αγοράς. Το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να πω είναι το τι γίνεται σε σχέση με τα λάθη. Κάθε μέρα βεβαίως με τις προτάσεις και στον προπολογισμό και οπουδήποτε βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει βεβαίως ε, και ε, ανοχή ε, και δεν είναι δυνατόν βεβαίως να κρύβουμε τα λάθη μας ε, αλλά ούτε και να κατηγορούμε την Κομισιόν όταν συμπεριφέρονται τσαπατσούλικα τα κράτη-μέλη με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. το πέρα αναφέρομαι στα διαρθρωτικά ταμεία. Αλλά Εγώ προσπάθησα κατά την διάρκεια της ε, θητείας μου να αλλάξω κάπως τα πράγματα. Πάλεψα ε, ήδη από το 2003 να υπάρξει κάπως μεγαλύτερη ευελιξία στον δημοσιονομικό κανονισμό ή σκεφτείτε το REACH παραδείγματος χάρη μια νομοθεσία μαμούθ. Ε, και εντάξει, Υπάρχουν βεβαίως κάποια λάθη και κάποιες λανθασμένες ε, υποθέσεις ε, ε, εργασίας. Δεν υπήρχε τότε η πολιτική βούληση να αντιμετωπιστούν αυτά. Ελπίζω να αλλάξει αυτό στην αναθεώρηση του ΡΙΤΣ. Βεβαίω. μην ξεχνάμε πως και αυτό θα ήθελα να συμβουλεύσω κάθε επίτροπο, πως θα πρέπει να, πρέπει να καταλάβουν όλοι οι υπαλλήλοι του το πολιτικό πνεύμα εντός του οποίου κινείται ο Επίτροπος. Να πω το εξής επίσης. Εγώ ήμουν στο διπλανό γραφείο με τον γενικό μου διευθυντή. Έτσι χτύπαγα την πόρτα και ερχόταν. Έχει μεγάλη σημασία αυτό στην Επιτροπή ε, πρώτη, που ήταν η πρώτη μου επιτροπή, καμιά φορά περνούσε μία εβδομάδα για να κλείσω ραντεβού με τον Γενικό Διευθυντή. Γιατί ε, εγώ ταξίδευα, εκείνο έλειπε, ήταν δύσκολα. Και θεωρώ πως η απόφαση να πάνε οι επίτροποι σε ένα κτίριο μακριά από την ε, γενική τους διεύθυνση θεωρώ πως είναι θεμελιωδώς ε, λανθασμένη. Εάν θέλει κανείς πολιτικό έλεγχο επί της υπηρεσίας, ε, πρέπει να βρίσκεται κανονικά και στο ίδιο κτίριο. Έχει σημασία αυτό. Τέλος. Βεβαίω είναι και ζήτημα ε, προσωπικότητας και του Επιτρόπου το εάν έχει ηγετικέ ικανότητες. Εάν έχει ηγετικές ικανότητες θα μπορέσει να διασφαλίσει την πρωτοκαθεδρία της πολιτικής. Εάν δεν τις έχει, εάν δεν θεωρεί εαυτόν ε, στοιχείο πολιτικής ηγεσίας αλλά την κορφή μιας διοίκησης, δεν θα είναι σε θέση να ασκήσει πολιτική ηγεσία και πολιτικό έλεγχο. Επί ενός ε, μηχανισμού ο οποίος είναι και σημαντικός και πραγματικά λειτουργεί σε... με πολύ ψηλές επιδόσεις. Σας Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα τα οποία μας είπατε. Ε, που προέρχονται βέβαια από την εμπειρία σας, τη μεγάλη εμπειρία σας. Βεβαίω θα έχουμε και την δυνατότητα να κάνουμε ερωτήσεις, αλλά τώρα θα ακούσουμε αμέσω τον κύριο Σεύκοβιτς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ο τίτλος της ομιλίας είναι «Το κόστος αποκέντρωση. Υπάρχει σαφής ε, διαχωριστική γραμμή μεταξύ πολιτικής και διοίκησης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνάδελφοι, καταρχά ευχαριστώ για την πρόσκληση για να συζητήσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γκρέσλε και τον Γκίντερ, αγαπητό συνάδελφο, για την εξαιρετική εισαγωγή του που μου επιτρέπει να επεκτείνω την παρουσίασή μου και σε άλλα θέματα. Διότι στην ουσία μιλάμε για αποκέντρωση, αλλά πολλά στοιχεία πρέπει να καλύψουμε. Η κυρία Γκρέσλερ αναφέρθηκε στα, στις διάφορες κανονιστικές υπηρεσίες της Επιτροπής που αναπτύχθηκαν ταχαίως τα τελευταία χρόνια και θα ασχοληθώ με το θέμα αυτό πριν το τέλος της παρουσίασής μου. Κατόπιν η δημιουργία εκτελεστικών οργανισμών που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Ενακτικό Συνέδριο για να βοηθήσει την Επιτροπή να εκτελέσει τα προγράμματά της με ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο και κατόπιν η δημιουργία διοικητικών γραφείων μέσα στην Επιτροπή που εξυπηρετούν και άλλους θεσμούς όπως ε, το Γραφείο Υποδομών εδώ και στο Λουξεμβούργο. Και εν τέλος θα ασχοληθώ και με το θέμα που ήδη αναφέρθηκε. Η αποκέντρωση από τις κεντρικές στις εξατομικευμένες υπηρεσίες, τις γενικές διευθύνσεις, τις διευθύνσεις και τα άτομα στην Επιτροπή. Κάτι που ισχύει για κάθε θεσμικό όργανο της Ένωσης νομίζω αντίστοιχα. Και εγώ θα συμφωνούσα με τον Κίντερ κάθε διεθνή διοίκηση. Το μεγαλύτερο τμήμα των ιδεών μου για τα θέματα αυτά είναι στο κείμενο που είχε προετοιμαστεί πριν τη συνάντησή μας και που νομίζω ότι περιλαμβάνεται στο βιβλιαράκι του Κοινοβουλίου. Επιτρέψτε μου λοιπόν να ακούσω τις συστάσεις της κυρίας Γκρέσλε να είμαι λίγο πιο αυθόρμητος και να μπω και σε άλλα θέματα που τέθηκαν από την προηγούμενη παρουσίαση. Πρώτον, η άποψη του πώς δουλεύει η Επιτροπή, τι όργανα, τι θεσμικό πλαίσιο χρειάζεται για την Επιτροπή. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε πολλά κοινά σημεία με τον κύριο Φεχόγγεν. Μην ξεχνάτε ότι η δουλειά της Επιτροπής και ο τρόπος λήψεως αποφάσεων καθοδηγείται από τη διασύνδεση μεταξύ των θεσμικών οργάνων, Επιτροπή Συμβουλίου και βεβαίως ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι λοιπόν η, κλασική σχέση που υπάρχει στα κράτη-μέλη, όπου η κυρίαρχη θεσμική σχέση είναι η σχέση πλειοψηφίας-μειοψηφίας του Εθνικό Κοινοβούλιο. Άλλο διακριτικό στοιχείο. Η Επιτροπή αποφασίζει με συλλογικό τρόπο. Πρέπει να υπάρξει συνένεση στο εσωτερικό της Επιτροπής και να προχωρήσουμε με πολύ δύσκολους, πολύ ειδικού φακέλους με επίγνωση του πνεύματος της συλλογικότητα. Και με έναν πολύ μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και αποφάσεις, γιατί συχνά οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεσμεύουν και μελλοντικέ επιτροπέ. Το Κοινοβούλιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσει, έντονες διαπραγματεύσεις για τα τελευταία στοιχεία του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου, που θα είναι ο προπολογισμό τη επομένη επταετία μέχρι το 2020. Είμαι βέβαιο λοιπόν ότι η επόμενη επιτροπή θα πρέπει να σεβαστεί τα ανώτατα όρια, τα επιμέρους ανώτατα όρια, όλες τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί εδώ και βέβαια υπάρχουν πολλές τέτοιες αποφάσεις που πρέπει να, να γίνουν σεβαστές και να τηρηθούν και από τα επόμενα εκτελεστικά όργανα της Ένωσης. Επίσης, έχουμε το ειδικό χαρακτηριστικό, είμαστε μια Ένωση 27 κρατών και οι αποφάσεις πρέπει να είναι αποδεκτές σε αυτούς. Θα έλεγα λοιπόν ότι η Επιτροπή και η Ένωση είναι μια δομή πολύ sui generis μοναδική ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά και είμαι πολύ προσεκτικός όταν κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ εθνικών κυβερνήσεων και επιτροπής. Υπάρχει βέβαια πάντα η συζήτηση για την πιο αποδοτική διοίκηση, για το πόσο γρήγορα οι πολιτικές αποφάσεις μπορούν να φτάσουν, να κατέβουν από τη γραφειοκρατία και να φτάσουν σε επίπεδο εκτέλεσης, υλοποίησης. Η προσωπική μου εμπειρία στην Επιτροπή αλλά και σε εθνικές δημόσιες διοικήσεις δεν θα σύστηνα το σύστημα κάτω από το οποίο με κάθε αλλαγή του κολεγίου να υπάρχουν ε, σημαντικές αλλαγές όλων, του όλων των επιπέδων της διοίκησης της Επιτροπής. Διότι ξέρω ότι αυτό θα οδηγήσει και οδηγεί σε πολλά κρατημέλη, σε απώλεια γνώση, σε απώλεια θεσμική μνήμης. Οι νέοι υπεύθυνοι χρειάζονται χρόνο να μπουν στο πετσί του ρόλου τους, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αν δουλεύουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να έχουμε επίγνωση της ανάγκης να μην δημιουργήσουμε καταστάσεις που θα οδηγήσουν σε εθνικά θέουδα συγκεκριμένων τομέων πολιτικής. Και ξέρετε πόσο σημαντική είναι η γεωγραφική ισορροπία για τα κράτη-μέλη, για όλα τα κράτη-μέλη και πόσο προσεκτικά παρακολουθούν τα νούμερα. Αν κατά πόσο δηλαδή η Ευρώπη, το ευρωπαϊκό πλαίσιο αντικατοπτρίζεται πιστά στη σύνθεση του προσωπικού των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Αν παρακολουθήσετε κάπως ε, τη διαδικασία των συστάσεων αναχώρα που εκδίδουμε κάθε χρόνο και εγώ τις παρουσίασα σε πολλά εθνικά κοινοβούλια, θα διαπιστώσετε νέα στοιχεία σε πολλά από αυτές τις συστάσεις. Η σύσταση για την ε, ικανότητα των εθνικών διοικήσεων. Είδαμε ότι σε πολλά κράτη-μέλη η διοικητική ικανότητα είναι συχνά ένας από τους λόγους γιατί δεν προχωρούν οι διαθροτικές αλλαγές, γιατί δεν υπάρχει ανάλωση των πόρων που επιμένετε, γιατί η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας πάει πιο πίσω από το χρονοδιάγραμμα. Εμείς συστήνουμε στα κράτη-μέλη αυτά να προσέχουν την νομοθεσία για τη δημόσια διοίκηση, την ανάγκη σταθερότητας, συνέχειας. Πιστεύουμε ότι τον 21ο αιώνα η διακυβέρνηση ενός κράτους είναι τόσο σύνθετη διαδικασία που πρέπει να έχει κάποιος καλούς επαγγελματίες για τη δουλειά αυτή. Βεβαίως, όπως τόνισε σωστά ο Γκίντερ, υπάρχουν ε, διαφορές, τριβές μεταξύ πολιτικού επίπεδου και διοίκηση. Και το ίδιο υπάρχει και στις εθνικές διοικήσεις, υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως τόνισε ο Γκίντερ, οι γενικοί διευθυντές είναι άτομα με μεγάλη εμπειρία, με ισχυρή προσωπικότητα. Χρειάστηκε να ακολουθήσουν ένα δύσκολο απαιτητικό ε, δρόμο και αποτελούν μια δυνατή προσωπικότητα. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι χρειάζονται ισχυρούς επιτρόπους. Πρέπει να υπάρχει μια συνεχής ε, αλληλεπίδραση μεταξύ τους για να διαμορφώνεται η πολιτική μέχρι τη λήψη της απόφασης. Και αυτό πρέπει να κρατάει λίγο. Βεβαίως η τελική απόφαση, αυτός που παίρνει την απόφαση, σε διαβεβαιώ ότι την παίρνει ο Επίτροπος και το Κολέγιο. Βέβαια, όσο μεγαλώνει το κολέγιο, όσο αποκτά περισσότερες ευθύνες, εξουσίες, κάτι που επεκτάθηκε σημαντικά πίν λόγω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της οικονομικής διακυβέρνησης. Η συλλογική προσέγγιση και η υποστήριξη προς τον πρόεδρο είναι κρίσιμου χαρακτήρα. Πρέπει επίση να ξέρουμε ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποστηριχθούν το Κοινοβούλιο. Δεν θέλουμε να υποβάλουμε προτάσεις χωρί να υπάρχει πιθανότητα να περάσουν. Γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε ούτε το δικό σα χρόνο, ούτε το χρόνο των κρατών μελών και θέλουμε αποτελέσματα. Όταν προτείνουμε κάτι λοιπόν, φροντίζουμε να περάσει από το κολέγιο, να τύχει υποστήριξη στο κοινοβούλιο και να γίνει δεκτό από τα κράτη-μέλη. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα γιατί ζούμε σε γρήγορες εποχές. Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται γρήγορα. Για το προσωπικό στην Επιτροπή δύο λόγια τώρα. Γιατί υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις και απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεται το προσωπικό της Επιτροπής και ποια είναι η σύνθεσή του. Ο μέσος όρος ηλικία όσων μπαίνουν στην Επιτροπή είναι τα 35 έτη. Η μεγάλη πλειοψηφία λοιπόν του προσωπικού της Επιτροπής είχαν μια προγενέστερη εμπειρία εκτός θεσμικών οργάνων ο καθηγητής κ. Κάσιν θα επιβεβαιώσει νομίζω ότι το προσωπικό της Επιτροπής έχει, είναι πολύ πολύ, σχηδές. Δεν είναι δικηγόροι η πλειοψηφία τους. Είναι οικονομολόγοι. Η δεύτερη δε ομάδα είναι οι επιστήμονες, δηλαδή η φυσική επιστήμη, η νομική είναι τρίτη. Μετά, σε ό,τι αφορά την ισορροπία φύλων τα τελευταία 30 χρόνια, το 2000, 46% του προσωπικού ήταν γυναίκες. Σήμερα είναι η πλειοψηφία, 53%. Μετά, χάρη στην πολύ καλή δουλειά του Γκίντερ Φεχόγγεν όταν ήταν επίτροπος διεύρυνσης, δεν έχουμε πλέον 15, αλλά 28 κράτη-μέλη στα θεσμικά κανά της Ένωσης. Για να υπάρξει λοιπόν, τον, όταν έχει κανείς την εντύπωση ότι είναι ένα κλειστό μαγαζί επιτροπή, χωρίς παράθυρα προς τον κόσμο, που δεν παίρνει νέα ρεύματα από τις διοικήσεις είναι λάθος. Μπορώ να σας πω ότι μέσα σε ένα σύστημα με τεράστιες αλλαγές στη, στα ανώτατα επίπεδα της διοίκησης υπάρχουν οι ίδιες δυναμικές αλλαγής και προσαρμογής στις νέες πραγματικότητες στην Ευρώπη. Αυτό που γίνεται στην Επιτροπή τα τελευταία 10-15 χρόνια. Ένα από τα προβλήματα που ανέφερε ο Γκίντερ είναι πώς θα κρατάμε τη δουλειά των Βρυξελών κοντά σε εσά, στους πολίτες, στις πόλεις. Πώς οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα επηρεάσουν την, την πραγματικότητα, την καθημερινότητα. Και εγώ είμαι από τους ισχυρότερους υποστηρικτές της διαφύλαξης των στενών σχέσεων με τις εξελίξεις στα κράτη-μέλη. Η διοίκηση της Ένωσης θα πρέπει, το πιστεύω αυτό, να αντικατοπτρίζει το ευρωπαϊκό τοπίο. Κάτι άλλο που θέλουμε να προχωρήσουμε, την εσωτερική κινητικότητα. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Επιτροπή ε, για χρόνια η νοοτροπία του ασύλου όπως τη λέγαμε. Δηλαδή κάνει κάποιος μια πρόταση, δεν, τη δια... δεν την ετοιμάζει με άλλους, μόνο μετά όταν πάει στην ε, ενδοϊπηρεσιακή διαβούλευση μπαίνει στη συζήτηση με άλλες δομές. Τώρα στην οικονομική διακυβέρνηση εισήχθη ένα νέο σύστημα που χρησιμοποιεί πολύ περισσότερο ένδο γενι... Ε, ε, ομάδες εργασίας μέσα στην ίδια γενική διεύθυνση μεταξύ γενικών διευθύνσεων που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτή την οτροπία ασύλου που βλέπουμε σε μεγάλο αριθμό εθνικών διοικήσεων. Μετά, σχέσεις με κράτη-μέλη και εμπειρογνωμοσύνη από τα κράτη-μέλη είναι παρόντα, πολύ έντονα παρόντα στην Επιτροπή. Έχουμε πάνω από χίλιους εθνικούς, αποσπασμέ, εθνικούς υπαλλήλους αποσπασμένους, έχουμε πολλούς ε, έκτακτους υπαλλήλους προσωρινής βάσης και κάνουμε και εξωτερική πρόσληψη ανα, αναπερίπτωση όταν θεωρούμε ότι χρειάζεται εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για το συγκεκριμένο θέμα. Ξέρω ότι το προσωπικό δεν το πολύ θέλει, ο κύριος Σεμπαστιάν ας πούμε, είχαμε κάτι έντονες συζητήσεις. Κάτι άλλο που θέλω να προτείνω και να ζητήσω την υποστήριξή σας για τις αθήκες εσάς. Η πρωτοβουλία που ανέλαβα για τη πρόθεσμη κινητικότητα μεταξύ Επιτροπής και Εθνικών Διοικήσεων και για τον ίδιο ακριβώ λόγο που ανέφερε ο Γκίντερ για να δει πώς θα φαίνεται η πραγματική ζωή. Βεβαίως, Χωρίς κώδικα διοντολογία τώρα είναι δύσκολο να έχουμε... Τώρα, τώρα με τον κώδικα διοντολογίας είναι δύσκολο να έχουμε υπαλλήλους, νέους υπαλλήλους να κάνουν στάσεις σε επιχειρήσεις. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε με εθνικές διοικήσεις. Και το λέω αυτό γιατί θεωρώ πολύ σημαντικό να ξέρουν οι υπάλληλοι μας ότι σε ένα μικρό φερρυπίν κράτο μέλος δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί μια σύνθετη νομοθεσία που υιοθετούμε. Είναι καλό να ξέρουν πώς οι εθνικές διοικήσεις αντιμετωπίζουν και δουλεύουν με τις ευρωπαϊκές απαντήσεις. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτό το κοινό πλαίσιο, το κοινό έργο της Ένωσης και η νομοθεσία που υιοθετούμε είναι κοινό στόχος και μπορεί να το πετύχουμε από κοινού. Συχνά, όταν μιλάμε για το μέγεθος της Επιτροπής, ακούει κανείς τον τύπο ότι, μιλάμε, ότι είναι μια τεράστια γραφειοκρατία με υπερπληθυσμό. Η Επιτροπή σήμερα έχει 30.000 προσωπικό περίπου. Βεβαίως μπορείτε να πείτε με ποιον το συγκρίνουμε. Εγώ είδα την διοίκηση της πόλης της Στοκχόλμης. Δεν θα σας εκπλήσει αυτό. Συμβαίνει αντίστοιχα σε πολλές άλλες πόλεις της Δυτικής Ευρώπης. Λοιπόν, η Στοκχόλμη έχει 40.000 υπαλλήλους. Θα μου πείτε βέβαια άλλες δουλειέ κάνουν. Έχουν άλλο ρόλο. Αλλά μιλάμε για μία πόλη από τη μια και για μία ήπειρο από την άλλη. Πόλεις σαν τη Στοχόλμη υπάρχουν πολλές στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 500 εκατομμύριων. Λάβετε υπόψη λοιπόν και τα μεγέθη αυτά. Τώρα αν συγκρίνουμε Υπουργεία και Γενικές Διευθύνσεις μπορείτε να κάνετε πολλές συγκρίσεις, δεν θέλω να σας ε, ζαλίσω με τα νούμερα. Δείτε δύο. Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών, MOVE, έχει προσωπικό 500 άτομα. Η MOVE. Δείτε το μέγεθος του Υπουργείου Μεταφορών της Βρετανίας. 1600 άτομα. Και επιπλέον έχουν και γραφεία ανά την Βρετανία και άλλα όπου έχουν άλλα 15.000 άτομα. Δεν κάνω παραλληλισμούς, απλά μεγέθη συγκρίνω. Δείτε τον τομέα της οικονομίας, όπου η Επιτροπή έχει περισσότερες εξουσίες και θα αποκτήσει περισσότερες ακόμα. Ας δούμε πόσο είναι το μέγεθος του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας. 1800 άτομα. Οι πιο συναφής διευθύνση οικονομικών, ECFIN, έχουν 1500 άτομα μαζί. Τι θέλω να πω. Με τις νέες ευθύνες της Επιτροπής, με τις νέες απαιτήσει γλώσσας, πρέπει να έχουμε 24 γλώσσες. Πρέπει να λειτουργούμε σε πολλές περιοχές, σε πολλές χώρες, σε πολλές περιφέρειες. Θα έλεγα ότι το μέγεθος της Επιτροπής δεν είναι εκτός πραγματικότητας. Προφανώς όμως μπορούμε να κάνουμε εξοικονομήσεις και θα σας τα πω όσον ούπο. Κάτι άλλο που και η κυρία Γκρέσλε και ο κύριος Φερχόγγεν ανέφεραν είναι τα πολιτικά χαρακτηριστικά των εθνικών ε, των, των 28 επιτρόπων. Όλοι λένε γιατί στις 28 περιορίστε τον αριθμό. Και πάλι αυτό που είναι σημαντικό να πούμε είναι δείτε το πολιτικό πλαίσιο των επιτρόπων. Είναι μόνοι τους. Δεν έχουν γενικούς γραμματείς, υφυπουργούς. Το πολιτικό πλαίσιο του κάθε επιτρόπου είναι ο ίδιος. Αν θέλετε λοιπόν, θες να συζητήσεις πολιτικά θέματα στην ε, Επιτροπή, στην ουσία πρέπει να πας στον ε, ε, Επίτροπο. Όχι λέει ο κ. Φερχόγγεν, πας στο Γενικό Διευθυντή. Όταν έχουμε εθνικά κοινοβούλια που θέλουν ε, να έχουν ακροάσεις για συγκεκριμένα ζητήματα, δεν θέλουν τον Γενικό Διευθυντή, θέλουν τον Επίτροπο. Αν πας στο Συμβούλιο Υπουργών, δεν πάει κανένας, ε, δεν γίνεται δεκτός κανένας πλην του Επιτρόπου. Και μετά υπάρχουν και οι διεθνείς υποχρεώσεις, η ομάδα των 8, η ομάδα των 20, ο ΠΟΕ. Δεν καθόμαστε. Αυτό θέλω να σας πω έχουμε πάρα πολλά σημαντικά ε, πάρα πολλές σημαντικές ευθύνες εκπροσώπησης και στους συνομοθέτες και σε διεθνές επίπεδο ενώ ταυτόχρονα πρέπει να καθοδηγήσεις και τις γενικές διευθύνσεις σου. Λάβετε και αυτό υπόψη όταν θέλετε να κάνετε συγκρίσεις με τις παραδοσιακές δομές των κρατών μελών. Έχεις υπουργούς, υφυπουργούς, μόνιμους γενικούς γραμματείς, γενικούς γραμματείς. Για μετρήστε τους. Θα εκπλαγείτε. Αποτελεσματικότητα τώρα. Ευχαριστώ και εδώ την Επιτροπή για τη στενή συνεργασία και τη συνεισφορά σας. Χάρη στη δουλειά σας και την αιμονή σας για τις εκθέσεις παρακολούθησης screening πολλά πράγματα στον τομέα. Ξέρετε ότι κλείσαμε τις διαπραγματεύσεις για το νέο κανονισμό του προσωπικού που θα ξεκινήσει του χρόνου τον Ιανουάριο, τον Ιανουάριο και θα έχει περικοπές αύξηση και θα εξοικονομήσει 2,5 δις. Πέραν αυτών που, είχε που είχαν εξοικονομήσει οι αλλαγές Κίνοκ το 2004 που από το 4 μέχρι το 20 είχαν 8 δισεκατομμύρια εξοικονόμηση. Οι συζητήσεις για τις περικοπές αυτές δεν ήταν εύκολες. Είχε ξεκινήσει πέρσι στην Επιτροπή. Δεν θέλω να σας πω πόσους καφέδες χρειάστηκε να πιω με τους συναδέλφους επιτρόπους για να βρούμε μια ισορροπία και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Ωστόσο βασίζουμε τις αποφάσεις μας στο screening. Μετράμε προσεκτικά τα overhead. Ε, μετράμε το workload της Επιτροπής και κάθε νέα έκθεση screening δίνεται από μένα πριν το κολέγιο, σε κάθε επίτροπο πριν γίνει συνέντευξη στο κολέγιο. Και έχω συζητήσει με τους γενικούς διευθυντές για το ποσοστό, τον αριθμό των αδειών ασθένειας, των αδειών, των ε, κενών ε, θέσεων. Όλα αυτά είναι χρήσιμα γιατί δείχνουν ότι Μπορούμε να πετύχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, να δούμε τα προβλήματα. Αυτό είναι ένα εργαλείο για το μέλλον. Γιατί τι θα γίνει την 1η Ιανουαρίου. Οι γενικέ διευθύνσει μπορεί μέσα στα επόμενα 5 χρόνια να χάσουν 10% του προσωπικού. 5% περικόπτονται και 5% μπαίνουν σε, αυτό το, ε, σε αυτή την ομάδα, την κοινή ομάδα κινητικότητας και δύσκολο, οδυνηρό εγχείρημα, αλλά με συγκεκριμένα νούμερα που πετύχαμε χάρη στο, στη διαδικασία screening. Μετά υπάρχει, υπάρχουν και άλλοι τομείς που μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Το ανέφερε ένα η κυρία Γκρέσλε. Απλοποίηση, καλύτερη διοίκηση. που μπορεί να γίνει με νέες τεχνολογίες. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη διαδικασία διεθνοποίηση. Πολύ δύσκολο. Είχα πάει στον Λευκό Οίκο να συζητήσω το θέμα αυτό με τον υπεύθυνο τεχνολογία του Λευκού Οίκου και τη ρώτησα ε, πώς το κάνετε εσείς αυτό και διαπίστωσα ότι απαιτείται IT, τεχνολογία πληροφορικής. Κάθε Υπουργείο Κάθε γενική διεύθυνση, στη δική μου περίπτωση, πρέπει να προσπαθεί να αναπτύξει το καλύτερο σύστημα της διεύθυνσης. Άρα τα συστήματα αναπτύσσονται με διαφορετικό τρόπο. Τώρα υπάρχουν περικοπές στον προπολογισμό, περικοπές στο προσωπικό. Άρα πρέπει να απλοποιήσουμε, να διευκολύνουμε τη διαδικασία και να έχουμε καλύτερο έλεγχο από ό,τι στο παρελθόν. Το ίδιο όταν προσφέρουμε υπηρεσίες από τη Γενική Διεύθυνση, επιτελικές υπηρεσίες, διότι στην πρώτη συνάντηση που είχε γίνει, ένα από τα συμπεράσματα στο οποίο είχαμε καταλήξει ήταν ότι όταν έχουμε συγκεντρωτισμό χρειάζεται, ε, χρειάζεται ισορροπία, ιδιαίτερα οι εταιρικέ υπηρεσίε, ανθρώπινοι πόροι, IT, που επιτρέπουν μείωση των overhead και επιτρέπουν στις γενικές διευθύνσεις να χρησιμοποιήσουν ε, περισσότερους πόρους για καλύτερους, τους ίδιους πόρους για περισσότερες δραστηριότητε. Εγώ μπορώ να σας πω ότι και καλό συντονισμό μπορεί να έχεις και καλή οργάνωση, στέρεη, ε, εταιρική ε, υποστήριξη στην Επιτροπή που θα επιτρέψει όλα τα θεσμικά όργανα να δουλέψουν καλύτερα. Να συνεχίσω για λίγη ώρα ακόμα. Αν για να την υποστήριξη σας στις κανονιστικές υπηρεσίες. Δουλεύουμε το θέμα αυτό και με την κυρία Γκρέστρε... και με άλλους συναδέλφους από το Κοινοβούλιο για χρόνια. Και μετά από τεράστιε προσπάθειες συμφωνήσαμε σε κάτι που πιστεύω ότι είναι μια οριζόντια προσέγγιση, πώς θα ρυθμίσουμε καλύτερα τις κανονιστικές υπηρεσίες. Έχουμε 49 υπηρεσίες αυτή τη στιγμή, 32 από αυτές έχουν κανονιστικό χαρακτήρα, είναι αποκεντρωμένα όργανα, ένας προϋπολογισμός 700 εκατομμύρια ευρώ και 7.000 και προσωπικό. Είναι καλό λοιπόν να υπάρξει σωστή διαχείριση και να υπάρχουν οριζόντιες αρχές που τις διέπουν. Προσπάθησα τις αρχές αυτές να τις εφαρμόσω από την πρώτη μέρα. Το πρώτο που ήρθε για διαπραγματεύση ήταν η υπηρεσία Σίπολ στη Βρετανία. Εγώ πρότεινα να συγχωνευτεί με τη Europol, διότι θεώρησα λογικό οι αστυνομικοί να καταρτίζονται κοντά στον βασικό στο βασικό όργανο της Ένωσης που ασχολείται με την αστυνομία. Επιπλέον η Βρετανική κυβέρνηση είχε πει σαφώ ότι θα μπορούσε να αφήσει την υπηρεσία αυτή να φύγει και θεωρήσε ότι είναι υπόδειγμα του τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, μέχρι το 2020 εξοικονομούμε 50 εκατομμύρια, χρησιμοποιούμε το προσωπικό της διοίκησης για ε, δράση και είναι ένα καλό, μια, καλή, μια καλή περίπτωση για να το χρησιμοποιήσουμε σαν παράδειγμα για μελλοντικές πίεσεις. Τι έγινε ούτε ένα κράτος μέλος, ούτε ένα, ούτε κι εσείς εδώ, υποστηρίξαν την συγχώνευση αυτή. Όλη η δουλειά που κάναμε λοιπόν δεν θα υλοποιηθεί όπως ελπίζαμε. Συχνά τα ίδια κράτη-μέλη και τα ίδια υπουργεία στα κράτη-μέλη που επικρίνουν επιτροπή λέγοντας περικόψτε, περικόψτε, περικόψτε, αλλάζουν άποψη για τη ΣΥΠΟΛ και τη Europol. Βοηθήστε με να το σπρώξω κάπως και να συζητήσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Γιατί αν δεν τα καταφέρουμε σε αυτό το σε αυτή την υποδειγματική περίπτωση, πολύ δύσκολο θα μπορέσουμε να κάνουμε ουσιαστικές συζητήσεις για άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες στο μέλλον. Ο, τώρα για να επανέλθω στον αρχικό τίτλο της ακροασής σας. Η Επιτροπή ως διαχειριστής του προπολογισμού. Είμαι πεπισμένος, και αυτό είναι πολύ χάρη και στη δουλειά της υπηρεσίας σας, ότι έχουμε τα σωστά εργαλεία, διαδικασίες, ελέγχους, για να εξασφαλίσουμε ότι ο προπολογισμό δαπανάται με τους κανόνες αποτελεσματικότητας που πρέπει και σε μερικές περιπτώσεις δίνουμε περισσότερο χρόνο για την τυπική συμμόρφωση παρά για τα αποτελέσματα, ουσιαστικά αποτελέσματα για τους πολίτες ή την κοινωνία. Το πώς θα βρούμε τώρα την ισορροπία αυτή απαιτεί μια καλύτερη διασύνδεση μεταξύ Επιτροπής και ημών. Το ελεγκτικό συνέδριο παίζει επίσης μεγάλο ρόλο, διότι πιστεύω ότι μόνο αυτή η στενή συνεργασία θα μας επιτρέψει να στείλουμε το σημαντικό αυτό μήνυμα που πρέπει να στείλουμε πριν τις επόμενες ευρωεκλογές μήνυμα ότι ο προπολογισμό της Ένωσης δαπανάται καλά. Ελέγχεται. Το 95% του προπολογισμού πηγαίνει, από τους, πηγαίνει στους πολίτες, στις περιφέρειες, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αυτό αποτελεί μια σημαντική επένδυση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δαπανώνται τα χρήματα ή υπό τους ενδεδειγμένους ελέγχους. Σας ευχαριστώ για την υπομονή, την καλή σας πρόσκληση και την ευγενική σας πρόκληση, πρόσκληση συγγνώμη, και την υπομονή να με ακούσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής. Ε, τώρα θα ακούσουμε δύο πολύ εξέχουσες προσωπικότητες ε, που παρακολούθησαν τις διαδικασίες μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κοιτάζω λίγο και το χρόνο. Έχουμε καθυστερήσει, αλλά πρέπει να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή. Οπότε, θα δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους για σύντομες ε, ε, ερωτήσεις, ε, δύο λεπτά. Πρώτα η κυρία Γκρέσλε, μετά ο κύριος Βαλτσίτης και δεν ξέρω ποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπατε και την σύναψη των όσων κάναμε τα τελευταία χρόνια. Εγώ θέλω να πω κάτι που δεν αναφέρθηκε. Ε, ένα πάρα πολύ σημαντικό φορέα εδώ πέρα. Την Γενική Γραμματεία και τι επιρροή έχει στους επιτρόπους. Νομίζω μπορείτε να μου πείτε κάποια πράγματα και εγώ ξέρω κάποιες ιστορίες. Εγώ βλέπω πως η Γενική Γραμματεία, παραδείγματος χάρη όταν μιλάμε για γραπτά ερωτήματα βουλευτών, ε, έχει πει πως οι απαντήσεις δεν πρέπει να είναι πάνω από 25 γραμμές. Και αναρωτιέμαι, πώς είναι δυνατόν να δέχεται ένα τέτοιο περιορισμό ένας επίτροπος. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν, γιατί το δέχεστε αυτό. Ευχαριστώ. Προτείνω να ακούσουμε πρώτα κάποιες ερωτήσεις και μετά. Σιγμάντας. Ačiū gerimas pirmininkė kadangi čia yra klausimai ir pasisakymai, aš daugiau norėjau pasisakyti šito klausimu. Pirmiausia, ευχαριστώ. Ε, ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Γκρέσλε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και μετά από τέσσερα χρόνια θητείας έχει φτάσει η ώρα αυτής της συζήτησης. Αλλά δεν ναι, μου φτάνουν δύο λεπτά και εμείς έχουμε μεγάλη εμπειρία και από το πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άλλοι ξέρουν το τι γίνεται στο Συμβούλιο. Γι' αυτό μπορώ να σας πω πως εγώ δεν μπορώ να πω πως ο ρόλος ε, του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου είναι αυτός που θα έπρεπε να είναι Έχουμε εγκρίνει πάρα πολλά μέτρα, π.χ. μηχανισμούς σταθερότητας και θεωρώ πως ο ρόλος του Επιτρόπου θα έπρεπε να επανεξεταστεί. Και συμφωνώ με την κυρία Γκρέσλε για το ρόλο της Γενικής Γραμματείας. Και θεωρώ πως ο ίδιος ο Επίτροπος πρέπει να είναι υπεύθυνο για τη δραστηριότητά του. Και εγώ είμαι υπέρ του να ξανασκεφτούμε πώς λειτουργεί το σύστημα γενικών διευθύνσεων και γενικής γραμματείας. Εάν δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να αντικαταστήσει ε, τον Γενικό Διευθυντή ε, επί σειρά ετών. Είναι πρόβλημα αυτό. Και θα ήθελα ε, να πω κάτι και στον κύριο Φερχόγγεν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να εξηγούν το τι συμβαίνει εντός της διοίκησης, εντός μιας ε, διεύθυνσης. Θεωρώ πως για το μέλλον θα ήταν σημαντικό η δραστηριότητα του κάθε επιτρόπου και του κάθε γενικού διευθυντή να αξιολογείται εδώ στο Κοινοβούλιο για να μπορούμε και εμείς οι βουλευτές να λέμε αν τα έχει καταφέρει στη δουλειά του ένας ε, γενικός διευθυντής ή ένας επίτροπος. Και, και οι εθνικές κυβερνήσεις λειτουργούν εν σώμα, θα έλεγε κανείς. Ψηφίζουν όταν υπάρχει διαφωνία και η πλειοψηφία αποφασίζει. Ε, ο χρόνος τώρα είναι περιορισμένος, δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά η σημαντικότερη μου σκέψη είναι εξής. Το θέμα αυτό της λογοθοσίας ε, ε, πρέπει να το ξαναδούμε για να μην έχουμε ξανά τέτοια ζητήματα όπως με την Όλαφ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάλι Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να μάθω τι γίνεται όντως με τη διάθεση των κονδυλίων εντός κομισιών. Σε ποιο βαθμό δηλαδή ο Επίτροπος μπορεί να εμπλακεί στην διάθεση των κονδυλίων. Για το θέμα είναι τι γίνεται στον έλεγχο και το τι εφαρμόζεται από αυτά τα οποία συμφωνούμε στον τριμερή διάλογο και το τι κάνουν βέβαια στα Εθνικά Υπουργεία στην εκτέλεση του προπολογισμού. Ευχαριστώ, δεν έχει δει κάποιο άλλο τον λόγο. Σίγμαν, θα σβήσει το μικρόφωνο σου, παρακαλώ. Ωραία. Μπορούμε να περάσουμε στι απαντήσει. Ο κ. Φερχόγγεν. Ευχαριστώ. Θα αναφερθώ πρώτα απ' όλα στο ερώτημα τη κυρία Γκρέσλε, γιατί είναι σημαντικό τα δέκα και μισό χρόνια που ήμουν επίτροπος, άλλαξε θεμελιωδώς ο ρόλος Γενικής Γραμματείας. Έζησα την εποχή Τρόγιαν, που θεωρούσε πως δουλειά του ήταν να τηρείται ο κανόνας της συλλογική λήψης αποφάσεων. Τυπικά δηλαδή έκανε τη δουλειά του. Ο διαδοχός του ήταν κάπως πολιτικός και μετά επί Μπαρόζο είχαμε τελείως πολιτικοποιημένη γενική γραμματεία η οποία τώρα είναι κατά κύριο λόγο θα έλεγα το εκτελεστικός κλάδος ε, του Προέδρου. Δηλαδή φροντίζει να επιβάλλεται η θέληση του Προέδρου της Επιτροπής να είναι ξεκάθαρο το τι επιθυμεί κτλ. Και υλοποιεί τις οδηγίες ε, του Πρόεδρου. Αυτό είναι το πρώτο. Μπορεί αυτό να σχετίζεται και με ε, προσωπικό ζήτημα, μπορεί να είναι και διαρθρωτικό, θα δούμε. Ο δεύτερος λόγος για το διαφορετικό ρόλο της Γενικής Γραμματείας είναι ε, η μεγαλύτερη ανάγκη συντονισμού λόγω αφενός της ε, διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέσω της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης. Και ενδιαφέρον είναι πως η Κομισιόν δεν το αγγίζει ευχάριστα αυτό το ζήτημα του εσωτερικού συντονισμού. Είχα συζητήσει και με τον Πρόντι και με τον Παρόζο για το πώς διασφαλίζει κανείς το ότι μία τόσο μεγάλη ε, κομισιόν ασκεί συνεπή ε, πολιτική και όχι κατακαιρματισμένη. Θα αναφέρω το παράδειγμα του Γερμανού διαδόχου μου, του Γκίντερ Έτιγκερ. Είναι σύμφωνα με το τίτλο αρμόδιος για την ενέργεια, αλλά αν το κοιτάξετε θα δείτε πως για ενέργεια είναι αρμόδιος και ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ανταγωνισμού, Κλίματος, Έρευνας, Εξωτερικού Εμπορίου κτλ. τα λοιπά, Και κανείς δεν συντονίζει το θέμα της ενέργειας εντός της Κομισιόν. Αυτός ο ρόλος λοιπόν ανήκει στη Γενική Γραμματεία. Και είναι πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Γιατί εκεί πέρα ακριβώς υπάρχει πολιτική συνοχή. Και μπορώ να σας πω κυρία Γκρέσλε. Οι περισσότερες αποφάσεις της Κομισιόν ε, λαμβάνονται χωρίς πολιτική συμμετοχή. Και δεν γίνεται αλλιώ. Είναι χιλιάδες οι επίσημες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν κάθε χρόνο. Υπάρχουν παραδείγματο χάρη εκατοντάδε περιπτώσει παραβιάσει τη συνθήκη. Θεωρείτε πω θα έχει διαβάσει ποτέ κανένα επίτροπο τι διαδικασίε αυτέ που κινούνται. Οι εκατοντάδε αυτέ αποφάσει λαμβάνονται χωρίς πολιτική ε, εμπλοκή των ε, επιτρόπων και είναι θέμα ακριβώς να διασφαλίζει ο Γενικός Διευθυντής μια πολιτική ε, συνοχή και γι' αυτό έχει γίνει τόσο σημαντική και ισχυρή Γενική Γραμματεία. Τώρα το τι μπορεί να γίνει, εγώ είμαι υπέρ της ε, ιδέας να είναι ξεχωριστή αρχή βεβαίως κομψιών, έτσι προβλέπουν οι συνθήκες, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μία αρχή χαρτοφυλακίων, με πολιτική ευθύνη και με διοικητική ευθύνη. Μετά, το ερώτημα του κυρίου Ρουμπιχ για τον προϋπολογισμό. Μπορώ να απαντήσω το, το πρώτο μέρος μόνο. Για το τι κάνει για την διάθεση των κονδυλίων ο Επίτροπος, τι επιρροή έχει. Μηδενική. Μηδενική ούτε επιρροή σε διαγωνισμό, ούτε σε απονομή συμβολέων. Και πρέπει να σου πω κύριε Ρούμπιχ, ευτυχώς, ευτυχώς κιόλας. Δεν χρειάζεται να σου πω πόσα τηλεφωνήματα δεχόμουν από περιφερειάρχες με αιτήματα, αν θέλετε, για να επηρεάσω τον προϋπολογισμό. Και τους έλεγα δεν μπορώ, δεν μπορώ. Όχι ότι δεν θέλω, δεν, δεν μπορούσα έτσι. Δεν μπορώ, δεν μου επιτρέπεται. Οπότε η επιρροή είναι μηδενική του Επιτρόπου. Και εδώ πέρα ακριβώς η απόφαση είναι των Γενικών Διευθυντών, οι οποίοι βεβαίως δεν ε, τρελαίνονται κιόλα. Δηλαδή ξέρω από το, τους δικούς μου γενικούς διευθυντές πως είχαν προβλήματα γιατί μετά υπάρχει και ζήτημα προσωπικής ευθύνης έτσι. Πρέπει να εξηγήσει ο άνθρωπος αυτός το γιατί έλαβε τη χύψη απόφαση. Και δεν τρελαίνονταν για αυτή την ευθύνη. Οπότε εδώ πέρα η Κομισιόν είναι πολύ, πολύ καλύτερα οργανωμένη από τις περισσότερες διοικήσεις που ξέρω. Γιατί η πολιτική επιρροή δεν είναι δυνατή από πλευράς εφαρμογής του προϋπολογισμού δηλαδή. Όσοι έχουμε λοιπόν κάποια εμπειρία από πολιτική, αυτό το θεωρούμε θετικό. Σας ευχαριστώ κύριε Φεχόγιν. Κύριε Σεύκοβιτς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ερωτήματά σας. Να ξεκινήσω με το Γενικό Γραμματέα, όπως είπε και ο Κούντερ. Υπάρχει και η εξουσία του Προέδρου που προέρχεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας και πρέπει να διαδραματίσει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Αυτό είναι προφανές και είναι γεγονός ότι οι μεγαλύτερες ε, ευθύνες ε, ε, της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, προέρχονται από την ανάγκη αναγκαίου συντονισμού. Και αυτό γιατί πρέπει να, γίνονται, να γίνεται συντονισμός κάποιων πολιτικών, ώστε δηλαδή μια πολιτική προερχόμενη από έναν τομέα να μην αντικρούει σε μια πολιτική από τον άλλο, να μην αντικρούει τον άλλον. Επομένως, πιστεύω ότι αυτός ο ρόλος συντονισμού είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δεν είναι μόνο γενικός γραμματέας ε, που το κάνει αυτό, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε πρέπει να γίνει από τα αρχικά στάδια των προτάσεων ο συντονισμό. και πρέπει οι πολιτικές ε, να παρουσιάζουν μια συνοχή όσον αφορά τώρα το ρόλο του Γενικού Γραμματέα μαζί με τον επικεφαλής ε, ε, της ομάδας του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλες αυτές οι συζητήσεις είναι συνήθως ε, μεγάλες συζητήσει, δύσκολες, προσπαθούν ε, να συγκεράσουν τις διαφορές και προσπαθούν ε, να δουν πώς θα λύσουν τα προβλήματα. Είτε μια συγκεκριμένη απόφαση ή είτε μια συζήτηση προσανατολισμού για το πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε κάποια πολιτική για το μέλλον. Ο Γενικός Γραμματέας είναι επίσης επικεφαλής ε, της ε, συνεδρίασης ε, των γενικών διευθυντών. Τους ενημερώνει για τα συμπεράσματα του Σώματος των Επιτρόπων και για το πολιτικό μέλλον. Εγώ έχω πολλές φορές συνεργαστεί με και έχω συμμετάσχει σε αυτές τις ε, συνεδριάσεις, απλώς και μόνο για να μπορέσω να πω στους συναδέλφους πώς ακριβώς, ε, βλέπουμε τον συντονισμό και τη συνεργασία με τον ε, Γενικό Γραμματέα και τους Γενικούς Διευθυντές. Όταν πρόκειται τώρα για τα συγκεκριμένα ερωτήματα προς βουλευτές, προφορικά ερωτήματα, το ερώτημα της κυρίας Γκρέσλε, είναι ένα θέμα που αφορά και τα εθνικά κοινοβούλια, γιατί υπάρχει, ε, ε, υπάρχει αίτημα για μεγαλύτερη ταχύτητα, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, για λεπτομερέστερες απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό. Γιατί αν ε, η πρόγνωσή μου ε, δεν είναι ε, λάθος, μπορεί 30.000 ερωτήματα να έχουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι κάνατε και έναν υπολογισμό του τι σημαίνει από απόψεως κόστους αυτό το κάθε ερώτημα δηλαδή του Ευρωβουλευτή, πρέπει να σας πω ότι πολλοί κόσμος δουλεύει για τα ερωτήματα αυτά των ε, ε, βουλευτών. Επομένως δεν υπάρχει καμία προσπάθεια ευθυγράμμισης με κάποιο γραφειοκρατικό τρόπο της απάντησης ε, την οποία δικαιούστε. Είναι γεγονός ότι αν είναι ευαίσθητο θέμα μπορεί να ξεπεράσει τις 25 σειρές και το βασικό ζήτημα είναι ότι πρέπει να δώσουμε κατευθυντήριες γραμμές ε, στους υπαλλήλους μας, πώς μπορούν να απαντήσουν, ποιος είναι ο συνήθις, ε, ποια είναι η συνήθις μορφή της απάντησης αυτή, αυτής. Ε, όταν τα ερωτήματα είναι από τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει, ε, χρειάστηκε να εισάγουμε ένα νέο σύστημα γιατί έχουμε και την κίτρινη κάρτα, έχουμε το θέμα της ελέγχου της επικουρικότητας, διαδικασία για την οποία πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ λεπτομερής, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να σεβαστούμε και τις προθεσμίες, οπότε έπρεπε να υπάρξει ένα νέο σύστημα ε, πληροφορικής για να, μπορέσουμε να μπορούμε να απαντούμε ε, στην ώρα μας. Αλλά να σας πω την αλήθεια, είναι πάρα πολλοί οι πόροι που χρειάζονται για κάτι τέτοιο ε, και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό πιο αποτελεσματικά. Βέβαια πρέπει να ασχοληθούμε και με τα ερωτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και με τα ερωτήματα από, το, τα Εθνικά Κοινοβούλια. Δεν ξέρω ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, ποια είναι η καλύτερη δυνατή λύση, γιατί υπάρχουν κάποια, κάποιες διαδικασίες ε, στην Bundestag για παράδειγμα, υπάρχουν κάποια όρια για τα ερωτήματα αυτά, για κάθε πολιτική ομάδα θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα ερωτήματα τα οποία ε, υποβάλλονται για παράδειγμα ε, που σκοπό έχουν απλώς ε, να ενισχύσουν τους, τις στατιστική για παράδειγμα να έχουν ίδιο χώρο στο σύστημά μας με καθαρά πολιτικού χαρακτήρα ερωτήσεις ώστε να μπορούμε να κάνουμε και εμείς καλύτερη δουλειά στην απάντηση των ερωτήσεων αυτών. Κύριε Μπαλτσίτης, ε, αναφερθήκατε στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στον Ευρωπαϊκό ε, Μηχανισμό σταθερότητας, όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την Ευρωζώνη. Φυσικά είναι ένα πολύ σημαντικό και ευαίσθητο θέμα. Και εδώ μάθαμε το μάθημά μας. Αν δεν μπορούμε να βρούμε μία λύση ε, βάσει του κοινοτικού ε, συστήματος και ε, μπούμε στον πειρασμό να ε, καλούμε εξωτερικούς εταίρους μας ε, στα του οίκου μας, στην καθαρά εσωτερική διαδικασία λήψη αποφάσεων αυτό, Σημαίνει ότι θολώνει κάπως η διαδικασία λήψης αποφάσεων και αυτό που υποφέρει περισσότερο είναι το ευρωπαϊκό όραμα, η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά και η κριτική ενάντια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ, πολύ ε, δρυμύτερη. Ελπίζω λοιπόν ότι από όλα αυτά θα μάθουμε για να ε, λειτουργήσουμε καλύτερα στο μέλλον. Πώς μπορούμε να, να... να βελτιώσουμε το συλλογικό περιβάλλον, με ρωτήσατε. Νομίζω ότι αυτό που θα περιμέναμε περισσότερο στο μέλλον ε, είναι μια καλύτερη, στενότερη συνεργασία ε, του Σώματος των Επιτρόπων. Όταν εγώ εκπροσώπησα την Επιτροπή στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων για πολλά χρόνια, ε, ήταν ένα από τα ερωτήματα που ετέθησαν από πολλούς. Πώς είναι δυνατόν ε, να συνεργαστούμε καλύτερα, ποια είναι ε, τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να το κάνουμε αυτό και όλα αυτά έχουν να κάνουν βέβαια και με τη συνολική μας την ευρύτερη την, την ευρύτερη πολιτική μας. Όσον αφορά τώρα το, τη συνεργασία και τον συντονισμό, ε, των Γενικών Διευθύνσεων, ε, των δραστηριοτήτων και του προπολογισμού. Ο κύριος Ρούμπικ έκανε αυτή την ερώτηση. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προσαρμοστεί στο νέο ρόλο και στις νέες, ε, στα νέα καθήκοντά της ως προς τον προϋπολογισμό να σας πω ένα παράδειγμα. Αν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος συνήθως είναι εκεί για να νομοθετεί, ε, λάβει ε, πολλά καθήκοντα και γίνει ξαφνικά υπεύθυνος για πάρα πολλά πράγματα, πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό το ρόλο του το εσωτερικό μας ε, σύστημα λογιστικού ελέγχου που εξασφαλίζει το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε ε, τα προβλήματα διαχείρισης ενός πολύ μεγαλύτερου προϋπολογισμού. Ε, τι γίνεται λοιπόν στις περισσότερες περιπτώσεις του συναδέλφου μου, τουλάχιστον, ετησί, τουλάχιστον εβδομαδιαίως έχουμε συζητήσει, συνεδριάσεις για να μπορέσουμε να παρουσιάζουμε τις, τα, τακτικά τις εκθέσεις δραστηριοτήτων, να δούμε πώς ακριβώς εκτελέστηκε προπολογισμό, αν υπάρχουν προβλήματα, αν υπάρχουν ατασταλίες ε, και έχουμε επίση και ένα πάρα πολύ καλό σύστημα εσωτερικού ελέγχου και εγώ είμαι τμήμα αυτής τη Επιτροπής ε, Εσωτερικού Ελέγχου, συμμετέχω σε αυτήν, τη οποία προεδρεύει ο Επίτροπος Σεμέτα ε, Όλοι λοιπόν, όλοι όσοι ε, έχουν αρμοδιότητα σχετική με τον προϋπολογισμό συμμετέχουν σε αυτές τις συνεδριάσεις. Είναι λοιπόν τμήμα της καθημερινής ε, ε, δουλειάς μας και φυσικά όλοι έχουμε μια προσωπική ευθύνη ε, όπως ε, και ε, οι γενικοί διευθυντές, οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το ρόλο τους αυτό και κάνουν ό,τι μπορούν για την καλύτερη εκτέλεση του προπολογισμού και να μην υπάρχουν ιδιαίτερα σφάλματα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο επιτρόπους για την παρουσίαση τους και για τις απαντήσεις στα ερωτήματα. Καθυστερήσαμε λίγο, αλλά θέλαμε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά με ανθρώπους που έχουν μεγάλη πείρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια να περιορίσει κανείς ε, τους ε, όσους προέρχονται από το πολιτικό φάσμα, αλλά ενδεχομένως οι επιστήμονες να τα καταφέρουν καλύτερα. Να ευχαριστήσω καταρχάς ε, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, ε, τον κύριο Σεύκοβιτς, αλλά και τον, ε, τον Κούτερ Φερχόγγεν, που ήταν πρώην μέλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και που παραστήκατε στην ακρόασή μας. Ja, dann darf ich als äh, nächsten Redner Herrn Stefan Becker von der Universität Speyer ganz herzlich hier begrüßen. Er wird zur Rolle des mittleren Managements. Ο κύριος Μπέκερ από το Πανεπιστήμιο Σπάιερ θα μας μιλήσετε για το ρόλο της, των μεσαίων στελεχών διοίκησης και του Γενικού Διευθυντή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν συντομότερο. Θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω μόνο 10 λεπτά από το χρόνο σα. Καταρχάς να σα ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μα δώσατε να ε, σα πούμε ποια είναι τα πορίσματά μας ε, για τα μεσαία και ανώτερα διοικητικά στελέχη. Ο συνάδελφο δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα. Θα σα παρουσιάσουμε λοιπόν μία εσωτερική θεώρηση των πραγμάτων, παρότι είμαστε ένα εξωτερικό παράγων. Ε, ελπίζουμε να μπορέσουμε να καλύψουμε τα θέματα της αποκέντρωσης, τη λογοδοσία και της αποτελεσματικότητας που είναι θέματα της σημερινή ακρόαση. Βασιζόμαστε σε πολλά ε, ερευνητικά προγράμματα της ε, των τελευταίων ετών. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο φάκελό σα. Πέντε προτάσεις θα σας προτείνουμε που πιστεύουμε ότι ε, καλύπτουν ε, τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μεσαία και ανώτερα στελέχη σήμερα. Η διοικητική μεταρρύθμιση δεν είχε τα αποτέλεσματα που περιμέναμε και μερικές φορές, όπως και αυτή τη φορά βέβαια, είχε κάποια απρόσμενα αρνητικά αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, έχει μία, ένα ακόμη κύκλο μεταρρύθμισης ε, που ε, δημιούργησε κάποια προβλήματα. Θα έπρεπε να έχει εξυγχρονιστεί κανονικά η διοίκηση ως προστατηγικό σχεδιασμό, την πολιτική για το προσωπικό και την οικονομική διαχείριση που μας ενδιαφέρει όλος ιδιωτόρο σήμερα. Για τα μεσαία και ανώτερα στελέχη, αυτό που θέλαμε ήταν, αυτό που ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ισχυθεί ο ρόλος της πρωτοβουλίας. Και αυτό σε κάποιο βαθμό έχει Αυτό που θέλαμε ε, είναι να υπάρχει υποστήριξη μεταξύ όσων αφορά κυρίως η μεταρρυθμίση αυτή, δηλαδή του προσωπικού. Τα ανώτερα στελέχη ήταν ιδιαίτερα επικριτικά στην αρχή, όμως σιγά σιγά η αντίθεσή τους αμβλήνθηκε γιατί ε, υπήρξαν παράλληλα και κάποιες εθνικές μεταρρυθμίσεις που υποβοήθησαν την όλη διαδικασία. Οι μεταρρυθμίσεις δεν ε, επιτυχάνουν πάντοτε 100% τους αρχικούς τους στόχους. Ε, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ε, υπάρχει πολύ μεγάλο διοικητικό άχθος σήμερα. Επίσης είναι αυτονόητο ότι η αποκέντρωση ε, έχει ως αποτέλεσμα και ένα επίπεδο ευξημένης λογοδοσίας και μερικές φορές δεν είναι πάρα πολύ καλή ισορροπία, όπως συμβαίνει και σήμερα, γιατί οι περισσότεροι γενικοί διευθυντές και τμηματάρχες λένε ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη γραφειοκρατία σήμερα, δηλαδή πολύ περισσότερα διοικητικά καθήκοντα και πιο σημαντικό ακόμα, πολλοί λένε ότι κάποια από αυτά τα νέα καθήκοντα είναι απλώς φορμαλιστικού χαρακτήρα, δηλαδή δεν έχουν πολύ αντίκτυπο στην καθημερινή σημερινή εργασία. Θα ήθελα να πω ορισμένα περισσότερα πράγματα ως προς αυτό, σε σχέση με το ρόλο των τμήματαρχών καταρχάς. Όταν αξιολογούμε το ρόλο τους, ο ρόλος που τώρα αξιολογούμε είναι σε σχέση με τον προηγούμενο τους ρόλους και αυτό βέβαια αφορά κυρίως ε, τα τμήματα ε, λήψη αποφάσεων για τις ε, διάφορες πολιτικές. Αρχικά οι τμήματάρχες ήταν καταρχάς υπεύθυνοι για την ανάπτυξη πολιτικής. Ήταν πολύ κοντά στο περιεχόμενο της πολιτικής και από την άλλη ήταν αρκετά υψηλά στην ιεραρχία για να μπορέσουν να συντονίσουν σωστά τα πράγματα. Τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι τα μεσαία στελέχη έχουν όλο και περισσότερα διοικητικά καθήκοντα, ειδικότερα ως προς το θέμα της διαχείρισης προσωπικού. Αυτό από τη μία σημαίνει ότι έχουν περισσότερη εξουσία σε σχέση με τους υφιστάμενους τους ε, ε, και έχουν λιγότερο χρόνο να φέρουν εις πέρα στα καθήκοντά τους. Δηλαδή αν δούμε ε, τους γενικούς διευθυντές, ουσιαστικά οι τμηματάρχες είναι αυτοί που σήκωσαν στους ώμους τους, στους ώμους τους το, την αλλαγή, ε, που, τη μεταρρύθμιση αυτή. Αυτό που παρατηρούμε επίσης είναι ότι υπάρχει μια αποξένωση μεταξύ του προηγούμενου ρόλου τους και την κατανόηση του ρόλου από τους τμηματάρχες ε, τους ίδιους, γιατί εξακολουθούν να θεωρούν ότι έχουν την πρωτοβουλία σε θέματα πολιτικής. Αυτό έχει σημασία για ολόκληρη τη μεταρρύθμιση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί ξέρετε ε, ότι ε, η μεταρρύθμιση όσο προχωράει ε, δυσκολεύουν τα πράγματα για όλο το προσωπικό. Ο καλύτερος τρόπος να πει κανείς, να συνοψίσει τη μεταρρύθμιση αυτή είναι η ενίσχυση του ρόλου του καθενός, το empowerment. Θέλησε δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πιο αυτόνομα τα διάφορα τμήματα ώστε ε, να μειωθούν, να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και για τους γενικούς διευθυντές, οι οποίοι έχουν τώρα μεγαλύτερη ευελιξία στην διάθεση των πόρων. Στην πράξη τώρα αυτό που βλέπουμε, και νομίζω ότι αυτό αναφέρθηκε ήδη και από τον κύριο Φερχόικεν, δεν θεωρούν ότι έχουν ενισχυθεί τα καθήκοντά τους, δεν αισθάνονται άνετα με την εξουσία που έχουν, για να το πω έτσι. Ε, υπάρχει το πρόβλημα του γραφειοκρατικού άχθους. Πολλές φορές ε, ισχυρίζονται ε, ότι έχουν όλο και περισσότερα πράγματα που πρέπει να ε, φέρουν εις πέρας. Πρέπει επίσης οι ανώτεροι, ε, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη να ελέγχουν τη δουλειά των υφισταμένων τους, κάτι το οποίο έχει ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό, ε, κάτι το οποίο ανέφερε και ο κύριος Φερχόγγεν. Οι περισσότεροι γενικοί διευθυντές θεωρούν ότι αυτό έχει παρατραβήξει. Ε, γιατί λένε ότι γνωρίζουν τους κινδύνους, κάτι το οποίο βεβαίως είναι καλό, αλλά οι περισσότεροι προσπαθούν να αποφύγουν όλους τους κινδύνους και αν ένας στόχος μεταρρύθμισης ήταν να ενισχύσει την ε, ε, πρωτοβουλία, πρέπει να σας πω ότι εδώ τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Όσον αφορά τώρα τις προηγούμενες ε, ε, αρμοδιότητές τους, ε, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα για τους γενικούς διευθυντές. Ένα ακόμη σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε σήμερα είναι η σχέση μεταξύ του πολιτικού και διοικητικού επίπεδου, δηλαδή μεταξύ του Επιτρόπου και του Γενικού Διευθυντή. Θα ακούσαμε και σήμερα ότι μπορεί να υπάρξει μεγάλη επιρροή όμως σήμερα ε, αναφέρεται ότι μπορεί να ισχύει μεν αυτό αλλά δεν θα πρέπει να ισχύει. Γιατί ε, κανένα ανώτερο τέλεχος δεν αντίκειται εσκεμένα στο, ε, στο πολιτικό επίπεδο. Στην πράξη όμως βλέπουμε ότι συμβαίνει αυτό και αρκετά συχνά και το είπε και ο κύριος Φερχόηγεν ότι αυτό έχει να κάνει με τον κάθε επίτροπο πόσο ο καθένας ε, αντιλαμβάνεται το ρόλο του. Κάποιοι είναι πιο δραστήριοι, έρχονται σε επαφή με το κάθε τμήμα τακτικά, άλλοι είναι κάποιο πιο παθητικοί και περιμένουν ε, ε, input από άλλους. Σε γενικές γραμμές ε, πρέπει να πω ότι ε, υπάρχει ικανοποίηση για τον τρόπο με τον οποίο ε, αλληλεπιδρά το διοικητικό με το πολιτικό επίπεδο και αν υπάρχουν κάποιες δυσκολίες είναι λογικό να ισχύουν αν το συγκρίνουμε και με το τι ισχύει στα εθνικά συστήματα. Ο συντονισμός τώρα μεταξύ των υπηρεσιών αναφέρθηκε προηγουμένως η γενική σοφία ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ κατακαιρματισμένη και ότι η διπηρεσιακή συνεργασία ε, δεν είναι ε, η κατάλληλη. Τα πορίσματά μας το επιβεβαίωσαν αυτό, αλλά υπάρχουν δύο στοιχεία. Πρώτον, τα μέσα και ανώτερα στελέχη ε, θεωρούν ότι είναι αποτελεσματική στο τμήμα τους η συνεργασία και η συνεργασία μεταξύ των τμήματων δεν είναι τόσο κακή όσο μερικές φορές αναφέρεται. Δεύτερον, δεν, ε, δεν είδαμε ότι δεν είδαμε να υπάρχει ε, μια σκέψη έτσι στενή με παροπίδες ε, σε γενικές γραμμές όλοι ασχολούνται με τις προεκτάσεις της πολιτικής με την οποία, για την οποία είναι υπεύθυνοι και ε, επομένως αυτή έτσι, η μεμονωμένη και απομονημένη θεώρηση των πραγμάτων ε, δεν ισχύει στο βαθμό ε, στον οποίο νομίζαμε. Βάσει των ευρημάτων αυτών προτείνουμε τις, τα εξής πεδία μετά από Πρώτον, όλα τα εργαλεία που εισήχθησαν κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων θα πρέπει να μπουν σε τεστ ε, λειτουργικότητας εμείς βλέπουμε ότι πολλά είναι δραστηριότητες που απλά επικυρώνουν κάτι. Δεύτερον, οι τμήματάρχες υφίστανται αυτή τη στιγμή μεγάλη γραφειοκρατική, πίεση. Άρα πρέπει να μειωθεί κάπως η πίεσή τους. Τρίτον, οι ανώτεροι, τα ανώτερα διευθυντικά στελέση έχουν μεγάλες ευθύνες οικονομική διαχείριση. Προτείνουμε επειδή υπάρχει κίνδυνος ε, προβλημάτων να μειωθεί. Τέταρτον, σχέσεις μεταξύ πολιτικού και διοικητικού επίπεδου. Χρειάζεται μια διευκρίνηση. Και σε άτυπο επίπεδο. Και πέμπτον, πρέπει να βελτιωθεί ο διυπηρεσιακός συντονισμός. Παρότι αυτό δεν είναι τόσο κακό, παρότι ο συντονισμός δεν είναι κακός, δεν είναι πολύ αποτελεσματικός. Αυτά είναι τα πέντε κύρια στοιχεία παρατηρήσεων μας για το ανώτατο, για το ανώτερο διοικητικό δυναμικό. Είμαι στη διάθεσή σας για απαντήσεις. Ευχαριστώ κύριε Μπέκερ. Τα είπατε λίγα και σταράτα. Θα τα συζητήσουμε μετά. Επόμενο θέμα, ο Χριστιανος Σεμπαστιάνη, πρόεδρος του της δομής του προσωπικού της Ένωσης θα μας δώσει την άποψη του προσωπικού για το θέμα της ε, αποκέντρωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού που επιβεβαίωσε την πρόσκληση πριν από πολλά χρόνια, το θύμισε η κυρία Γκρέσλε. Δεν ξέρω αν αυτοί που κέρδισαν ήταν οι γενικοί διευθυντές, αυτοί που χάσαν είναι πολλοί και είμαι εδώ για να προσπαθήσω να κάνω όχι μόνο τον απολογισμό του τι είχε γίνει πριν από 10 χρόνια, αλλά να δούμε τι θα μπορούσε να είχε γίνει για να βελτιώσει τις, ε, τα αρνητικά, διαπιστώσεις. Πριν μπω στην ουσία του θέματος, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω στο, εσάς του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής του Ελέγχου Προϋπολογισμού, γιατί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη μεταρρύθμιση ήσασταν κριτικοί χωρίς να είσαστε καταστροφικοί. Είχατε ε, στόχο τη διατήρηξη των βασικών ε, θέσεων της ε, Ευρωπαϊκής Δημόσιας Διοίκησης και ευχαριστώ την Αντιπρόεδρο που ήταν υπέρ της επικεφαλής διαπραγμάτευσης. Εμείς είμαστε υπέρ των εισαγωγών που κάνατε, ιδιαίτερα ότι αφορά τις, τις, τις συμφερόντων, Η μελέτη που παρουσιάζεται είναι πολύ διαυγής. Ε, η μεταρρύθμιση δεν ξεκίνησε από την ανάλυση της βελτίωσης ε, της ε, αποτελεσματικότητας αλλά από την προάσπιση της λογοδοσίας. Δηλαδή στηριζόταν στην ευθύνη αλλά όχι στη λογοδοσία. Ενώπιον της διαπίστωσης ότι δεν μπορούσαν να ελεγχθούν τα πάντα, η περιορίστηκε σε μια λογική ε, στεγανών όπου ο καθένας είναι υπεύθυνο για τα δικά του αλλά κανείς δεν υπεύθυνο για όλο το θεσμικό πλαίσιο. Στην τελευταία ακρόαση θυμάμαι ένα επεισόδιο που είχαμε τον κύριο Κλοντσέν, Γενικό Διευθυντή Διοίκηση τότε, που σε μία απάντηση σε ερώτηση, τη απαντήσει της Γκρέσλε ότι ήταν αδύνατον να πιστεύει ότι η Κομισιόν ήταν ένα όργανο, αν έβλεπε κανείς μόνο το, το οργανόγραμμα της Επιτροπής και είχε πει ε, ότι αν πάω να κάνω κάτι τέτοιο θα μου την πέσουν ή ε, του προσωπικού. Εμείς συμβάλαμε ωστόσο στην ε, θετική μεταρρύθμιση γιατί συμμεριζόμαστε το πνεύμα που την διέπε. Η διαπίστωση της κρίσης ήταν η παρεκκλήση στους πιο αποκεντρωμένους τομείς ε, που ήταν ο τομέας της έρευνας όπου υπήρχε σαφής έλλειψη ε, συντονισμού σε τοπικό επίπεδο η απάντηση θα φανταζόταν κανείς είναι καλύτερος συντονισμός. Διαπιστώνουμε μαζί ότι δεν ήταν αυτή η απάντηση. Η, ανταλλαγή, η αλλαγή αυτή η προσέγγιση είχε αντίκτυπο και στην αντίληψη που είχε κάθε υπάλληλο για το ρόλο του. Περάσαμε από τη λογική της ε, ταυτάφτισης της νομιμοφροσύνης προς την Επιτροπή, αυτός που επιλέγει την υπηρεσία δεν παραμένει υπεύθυνος και πέραν του ορίου παραγραφής. Τώρα έχουμε μετατραπεί σε μια μισθοφορική νομιμοφροσύνη προς τον επικεφαλή σου. κ. Φερχόγγεν ε, περιέγραψε καλά το ρόλο των μεγαλομανών ε, νέων υπαλλήλων που νομίζουν ότι αυτή είναι η επιτροπή. Καρικατούρα μεν, αλλά βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ε, υπάρχει η τάση να προσπαθείς να κάνεις καριέρα μέσα στον χώρο σου και δεν υπάρχει εικόνα της ενότητας ε, της, ε, των υπαλλήλων της Επιτροπής εξού και η έλλειψη εμπιστοσύνη των πολιτών. Δεν καταλαβαίνουν την ταυτότητα της Επιτροπής, έχουν μπροστά μια σειρά στεγανών ανεξάρτητων μεταξύ τους. Γιατί η σύγκρουση μεταξύ Φερχόγγιν και Γενικού Διευθυντού του ήταν ε, διαφορά για το ποιος είχε, έκανε κουμάντο. Αλλά και οι δεύτεροι θεωρούσαν ότι δεν ήθελαν να ακούσουν τις απόψεις Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων ή του, της Γενικής Αυτό σημαίνει μεγάλη απώλεια πόρων και εξαιρετική έλλειψη αποτελεσματικότητας. Αυτό που είχε γίνει μετά την τελευταία συνάντησή μας δεν είναι τόσο αρνητικό πάντα γιατί μπορεί να ρωτήσει κανείς υπήρχε μια επίγνωση. Η αποκέντρωση των εκτελεστικών κανονιστικών υπηρεσιών ήταν αποτέλεσμα της ίδιας αντίδρασης. Ε, εκχωρούμε αρμοδιότητες που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα ιδίω για να μην έχουμε ευθύνη αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα ιδίω έναντι του Κοινοβουλίου τη Επιτροπή Ελέγχου του προπολογισμού. Είχα συνοδεύσει τον κύριο Κάλλα σε μια συνάντηση με εκπροσώπους του προσωπικού των ε, κανονιστικών υπηρεσιών και σαν αστείο τους έλεγε είμαι βέβαιο ότι θα πάω κάποια στιγμή στην Κοκομπή γιατί κάποιος παλαβός ε, διευθυντή αγόρασε χρυσέ μπανιέρες. Εγώ θα φροντίσω αυτό να μην γίνει και είμαι εδώ για να σας βοηθήσω γι' αυτό, έλεγε ο κύριος Κάλλας, να ελέγξουμε και να επαγρυπνούμε πάνω στις δαπάνε. Έκτοτε έγιναν πολλά πράγματα, δεν θα αρχίσω να επενώ την Επιτροπή, που κάνουν όλοι οι Επιτροποί, αλλά μπορώ να σας πω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της μεταρρυθμίσης του καταστατικού που έχει πολύ καλύτερους κανονισμούς λειτουργίας του προσωπικού, για το προσωπικό των υπηρεσιών, υπάρχει εναρμόνιση κανόνων, υπάρχει μητρό καταγραφής του τρόπου εφαρμογής του καταστατικού για να μην υπάρχουν αποκλίνωσες εφαρμογές και ε, η Επιτροπή αντιλήφθηκε ότι η αποκέντρωση δεν είναι η λύση. Αρχίζει λοιπόν να επανασυγκεντρώνει και είμαι εδώ για να σας πω και άλλα καλά νέα. Παραδείγματος χάρη στον τομέα της έρευνας όπου είχαμε εκτελεστικές ε, υπηρεσίες μετά από σχέδιο απόφασης επιτροπής ε, του κ. Σεύκοβιτς και Λεβαντόφσκι ε, περιλαμβάνονται ενδιαφέρουσες ιδέες για το προσωπικό. Πέντε κεντρικές υπηρεσίες. Δεν θα υπάρχουν οι πολλαπλές νομικές ερμηνείες των ίδιων κανόνων στη διαχείριση της έρευνας. Μία κεντρική υπηρεσία ελέγχων, μία κεντρική υπηρεσία IT, μία κεντρική υπηρεσία διάδοσης της πληροφορίας είναι προγράμματα έρευνας προς όφελος των δικαιούχων. Δεν μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές εφαρμογές στους κανόνες. Και εγώ ασχολούμαι στη γενική μου διεύθυνση με τις κρατικές αγορές. Το πρώτο μου ερώτημα που μου λένε είναι η διπλανή γενική διεύθυνση κάνει το ανάποδο. Τι μας λέτε ότι είστε το ίδιο όργανο. Και επιπλέον προτείνεται ένα steering committee όπου οι κεντρικές υπηρεσίες παρίστανται, εκπροσωπούνται και που αποφασίζει, απο, λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία. Ε, πρόκειται για τελείως διαφορετική προσέγγιση. Ελπίζω το σχέδιο αυτό να υλοποιηθεί, γιατί πραγματικά θεωρούμε, τουλάχιστον εμείς, ότι πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν προχωρήσουμε τώρα στις κανονιστικές υπηρεσίες, βλέπουμε σοβαρή έλλειψη συντονισμού για την συμμετοχή εκπροσώπων της Επιτροπής. Ε, στέλναμε ειδικού στους τομείς δραστηριότητας της Ένωσης που δεν είχαν γνώσεις ή αρμοδιότητες για τους κανόνες διαχείρισης προσωπικού και διοίκησης. Πρόκειται για πρόβλημα της Γενικής Γραμματείας που από ό,τι φαίνεται καλύπτεται σιγά σιγά διότι η Επιτροπή συντονίζει περισσότερο το, τα μέλη στα ε, στις, ε, στα διοικητικά συμβούλια. Σε κάθε περίπτωση έχει δικαίωμα βέτο. Πρέπει να χρησιμοποιεί το δικαίωμα αυτό για να μπλοκάρει αποφάσεις που λαμβάνονται από άτομα που δεν έχουν την ικανότητα ούτε την ευαισθησία της ε, Ευρωπαϊκής Δημόσιας Υπηρεσίας και προσπαθούν να περάσουν θέσεις τους. Αυτά είναι μηνύματα που πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Εμείς επικρίνουμε αλλά προσέχουμε και τις ε, εξελίξεις και είμαστε εδώ για να ενισχύουμε γιατί επιλέξαμε να υπηρετήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουμε να ανήκουμε σε μία γενική ε, διεύθυνση, σε έναν κλάδο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε καλύτερα την δομή της ε, υπηρεσίας, να λάβουμε υπόψη τον πολίτη και να μην τσακωνόμαστε για το ποιο θα είναι το αφεντικό ενός μικρού απομονωμένου νησιού. Δεν είναι η φεουδαρχική εποχή. Σήμερα είμαστε στην εποχή της δημοκρατίας. Όλοι ξέρουμε ότι λειτουργούμε στα πλαίσια ενός θεσμικού οργάνου, όχι ως άτομα. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε υπεύθυνοι, εργαζόμενοι μιας υπηρεσίας. Όπως ξέρετε οι περισσότερες δράσεις περιλαμβάνονται ε, στις δράσεις, στις δραστηριότητες επαγρύπνησης. Εμείς θεωρούμε ότι ο οργανισμός μας πρέπει να μπορεί να αλλάξει μόνος του, όχι να μας τον επιβάλλουν συνεχώς ε, οι άλλοι. Που με κριτικές δεν ακολουθούν πάντα, δεν έχουν πάντα ως στόχο την ε, βελτίωση της υπηρεσίας, αλλά και άλλους στόχους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σεμπαστιανή για αυτά τα οποία μας είπατε από την πλευρά του προσωπικού. Μιλήσατε για ζήτημα αποκέντρωσης ε, και για το εάν αυτή προχωράει ή όχι. Θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε κατόπιν στην βίλε, του Πανεπιστημίου του Λάιντεν για την ανάγκη που υπάρχει να υπάρξει αποτελεσματικός έλεγχος από πλευράς ε, Κοινοβουλίου. Καλώς ήρθατε κυρία Βίλε. Τι αποτελέσματα λοιπόν είχε η αποκέντρωση στην δυνατότητα του Κοινοβουλίου να ελέγχει πλήρως ε, την εκτελεστική πτυχή. Ήθελα λοιπόν να σας δώσω αμέσως ε, τον ε, λόγο. Δουλεύει το μηχάνημα να μας δείξετε αυτά που θέλετε. Όχι. Έχετε λοιπόν το λόγο. Εντάξει. Τέλο πάντων, αν δεν μπορείτε να τη δείτε τι διαφάνειε, είναι στο φυλάδιο που σα έχω δώσει. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση να παρευρεθώ στην ακρόαση αυτή. Εγώ το είδα λίγο στενά το θέμα, δηλαδή ότι έπρεπε να εστιάσω στην οικονομική λογοδοσία εντός της ε, Κομισιόν. Η δε συγγήτρια μου είπε να το δω λίγο ευρύτερα. Θα προσπαθήσω με βάση τα ευρήματα της μελέτης ε, που δημοσίευσα το καλοκαίρι με βάση το βιβλίο μου που εξέδωσε το Πανεπιστήμιο της ε, Οξφόρδης. Κοιτάξτε, έχω πρόβλημα με τις φωνητικές μου χορδές, οπότε καμιά φορά η φωνή μου ακούγεται σαν να τρέμει. Αλλά ε, πέρα από τη συγκίνηση βεβαίως ε, δεν, δεν κλαίω. Κάποια νευράκια έχω, αλλά τέλος πάντων δεν είναι το θέμα μας αυτό. Θα προσπαθήσω πρώτα απ' όλα να πω λίγα λόγια για τη λογοδοσία. Γιατί είναι μια λέξη πολύ της μόδας ε, τελευταία ειδικά βεβαίως σε ρητορικά σχήματα πριν ε, προχωρήσουμε ας δούμε τον ορισμό της ε, λογοδοσίας σημαίνει πως οι υπάλληλοι θα πρέπει να αποκαλύπτουν πληροφορίες για να εξηγούν τι, πώς ασκούν την εξουσία που έχουν. Οπότε υπάρχουν τέσσερα στοιχεία. Πρώτον, κάποιος ο οποίος θα λογοδοτεί, άνθρωπος ή θεσμικό όργανο. Ένας τομέας αρμοδιοτήτων. Η ύπαρξη ενός βήματος λογοδοσίας ε, μπορεί να είναι π.χ. το κοινοβούλιο, μπορεί να είναι πολιτικό, διοικητικό, νομικό και το δικαίωμα αυτού ο οποίος ελέγχει να ενημερώνεται, να κρίνει και να επιβάλλει κυρώσεις. Δηλαδή, με λίγα λόγια θα λέγαμε ποιος είναι υπόλογος, γιατί, σε ποιον και πώς, με ποιο τρόπο. Συχνά λοιπόν η λογοδοσία σημαίνει πως ε, θα πρέπει βεβαίως να αναμένουν ότι θα δώσουν λόγο η τα μέλη της διοίκησης, αλλά βεβαίως και υπάρχει ο εξπόστ έλεγχος. Τι βλέπουμε λοιπόν από τη μελέτη που κάναμε είναι πως υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανισμοί λογοδοσία εντός και γύρω από την Κομισιόν. Είχαμε βεβαίως την παρέτηση της Επιτροπής Σαντέρ που έπαιξε ρόλο καταλητικό και αυτό σημαίνει πως πολλές εσωτερικές διοικητικές μεταρρυθμίσεις ε, που μετασχημάτισαν την Κομισιόν αλλά ταυτόχρονα είχαμε και κάποιες ε, πολιτικές τέτοιες μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν τη λειτουργία της Κομισιόν. Και βέβαια ε, αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τον εξυγχρονισμό του μηχανισμού λογοδοσίας. Βλέπετε τις ε, λεγόμενες προεδρικές εξουσίες, ε, τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές και τον κώδικα συμπεριφορά. Εσωτερικά υπάρχει ε, ένας προγραμματικός κύκλος στρατηγικού σχεδιασμού και ένα σύστημα οικονομικής λογοδοσίας που ήταν η βασική μορφή του μετασχηματισμού στο επιχειρησιακό επίπεδο. Μετά, Αυτά βεβαίως δεν περιορίστηκαν σε εσωτερικές αλλαγές αλλά και σε εξωτερικές. Μπορώ μάλιστα να πω πως εξωτερικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, είχε επέκταση του ρόλου του όσον αφορά τους ελέγχους ex post επί της Κομισιόν και εξάντε και ταυτόχρονα στον διοικητικό τομέα βλέπουμε την ε, ισχυροποίηση του ελεγκτικού συνεδρίου του διαμεσολαβητή και του Όλαφ. Οπότε έχουμε αυτές τις... και την πρωτοβουλία διαφάνειας βεβαίως. Οπότε είχαμε βεβαίως και τα της ε, λογοδοσίες η οποία κατέστη ένα φυσιολογικό μέρος της λειτουργίας της ε, Κομισιόν. Τα επανέλθω αυτό αργότερα. Τώρα θα μείνω λίγο στη λογοδοσία στα ζητήματα τα οικονομικά. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες που βλέπετε στη διαφάνεια. Να πω μόνο πως η λογοδοσία στον οικονομικό τομέα δεν είναι κάτι που γίνεται άπαξ με μία μεταρρύθμιση, αλλά είναι ένα πακέτο ευρύτερων μεταρρυθμίσεων. Π.χ. στην Κομισιόν βλέπουμε πως η ευθύνη των υπηρεσιών με τις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις ΚΙΝΟΚ κατέληξαν σε μια πιο αποκεντρωμένη ε, χρηματοοικονομική διαχείριση και βεβαίως ε, στο επίπεδο διευθυντού, γενικού διευθυντή και μέσης διοίκησης υπάρχει η αίσθηση της ευθύνης για τα οικονομικά. Και βέβαια αυτό ε, γίνεται και με την σύσταση μιας υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο τμήματος και με την κεντρική βεβαίως ε, υπηρεσία της Κομισιόν, κάτι το οποίο σημαίνει κάποια επαγγελματική ε, στήριξη και βεβαίως υπάρχουν και μεταθέσεις από τις ε, ευαίσθητες ε, θέσεις ε, κάθε επταετία και βεβαίως υπάρχουν και οι αλλαγές στην συνθήκη που κατέστησαν την Κομισιόν μια πιο φυσιολογική εκτελεστική διοίκηση. Ας δούμε λίγο την διοίκηση και την δομή της οικονομικής λογοδοσίας, πλέον είναι σαφές ποιος είναι υπεύθυνο για την διαχείριση. Αυτό σημαίνει πως τα υψηλόβαθμα στελέχη κινητοποιήθηκαν όσον αφορά την διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων των τμήματων τους. Υπάρχει η έμφαση της ατομικής ευθύνης του Γενικού Διευθυντή. Τα υψηλόβαθμα στελέχη προσωπικά α, πρέπει να και επομίζονται τις συνέπειες της απόδοσής τους. Πώς γίνεται αυτό. Έχουμε την ετήσια έκθεση αναφορών που πρέπει να υποβάλει ο Γενικός Διευθυντής ε, και δίνει λόγο για το πώς διαχειρίστηκε τους πόρους του, ε, τις δηλώσεις και βεβαίως και ε, τα σημεία στα οποία υπάρχουν τυχόν επιφυλάξεις εντό της έκθεσης λίγο Αν δούμε λοιπόν το τι είναι το αντικείμενο του ελέγχου. Υπάρχει μια σαφής διάκριση μεταξύ του πολιτικού και του διοικητικού επίπεδου. Επίτροποι και γενικοί διευθυντές έχουν τομείς ευθύνης που αλληλεπικαλύπτονται όπως βλέπετε ως ένα βαθμό. Βλέπετε στο σχήμα. Και αυτό είναι βεβαίως κάπως αναπόφευκτο σε μια διοίκηση όπως Κομισιόν, όπως και στις εθνικές διοικήσεις, αλλά πολύ περισσότερο από ποτέ υπάρχουν, υπάρχει σαφής διάκριση των αρμοδιοτήτων, επιτρόπων, πολιτικών, δηλαδή και των γενικών διευθυντών. Ναι, υπάρχει αμφιβολία πως η σαφεστρευτή διάκριση σχετίζεται με τον ισχυρότερο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. από πλευρά νομοθετικών αρμοδιοτήτων που σημαίνει πως ε, ο Επίτροπος έχει πολιτική ευθύνη η οποία βεβαίως συνδέεται με την ευθύνη του Γενικού Διευθυντή. Τι είναι λοιπόν σημαντικό δεν είναι μόνο οι νέες μορφές λογοδοσίας και διατάξεις, κυρώσεις κτλ. Αλλά επίσης το ότι υπάρχει ε, ένας ε, νομοθέτης, ένα νομοθετικό σώμα που ε, ασκεί έλεγχο επί του εκτελεστικού. Και εδώ πέρα πλέον είναι πιο ξεκάθαρος ο διαχωρισμός ε, και πολιτικής. Επίσης βλέπουμε πως υπάρχει και μια σαφής ιεραρχική σχέση μεταξύ πολιτικής και διοίκησης, κατά το οποίο συλλογικό. Γιατί βεβαίως στη βιβλιογραφία τη σχετική ε, αναφερόμαστε στον Μαξ Βέμπερ ο οποίος ε, μίλησε για κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ πολιτικής και ε, πολιτικών και διοίκησης. Έχει συγγράψει σημαντικά έργα και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι πως πλησιάζει στο βεμπεριανό μοντέλο η Κομισιόν. Βλέπουμε τον ισχυμένο ρόλο του Κοινοβουλίου ως το μέρος όπου ασκείται η λογοδοσία. Γι' αυτό λέω πως δεν είναι μόνο εσωτερική η διαδικασία, Είχαμε και τις μεταρρυθμίσεις της ε, συνθήκης που βεβαίω επέβαλαν την αρμοδιότητα αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την εσωτερική λειτουργία της Κομισιόν. Υπάρχει λοιπόν ισχυρότερος πολιτικός έλεγχος επί της Κομισιόν. Έχουμε και τον ρόλο του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και τις κατευθυντήριες γραμμές και τις πενταετής κατευθυντήριες γραμμές και βλέπουμε βεβαίω το τι γίνεται από πλευράς λογοδοσίες. Υπάρχει επίσης αποπολιτικοποίηση της διοίκησης Περισσότερη έμφαση δίνεται στην απόδοση, στον επαγγελματισμό, στην ευθύνη και οι διαδικασίες πρόσληψης επίσης αποπολιτικοποιήθηκαν και αποεθνικοποιήθηκαν. Γιατί η αποεθνικοποίηση ε, ήταν πάρα πολύ σημαντική και στο διοικητικό επίπεδο και πλέον υπάρχει ξεκάθαρη διαφοροποίηση πολιτικών και διοικητικών σφαιρών. Υπάρχουν λοιπόν δύο τάσεις που είναι ορατές. Πρώτα απ' όλα ένας διαχωρισμός όσον αφορά τις ευθύνες, όσον αφορά τις προσλήψεις, δηλαδή οι επίτροποι οι ίδιοι έχουν καταστεί πιο πολιτικά πρόσωπα οπωσδήποτε και η ε, κορυφή της διοίκησης έχει αποπολιτικοποιηθεί. Αυτό φαίνεται και στο, στον τομέα των ευθυνών και το, της πολιτικής προσωπικού αλλά και στις προσδοκίες Δηλαδή αυτό το οποίο αναμένεται από τον Επίτροπο είναι ένας πολιτικός ρόλος και αυτό το ακούσαμε μόλις και αυτό το οποίο αναμένουμε από την κορυφή της διοίκησης είναι να είναι διαχειριστές. Έχουμε λοιπόν μία τάση που είναι ο διαχωρισμός. Το άλλο είναι μία ιεραρχική σχέση. Υπάρχει λοιπόν μια βεμπεροποίηση θα λέγαμε. Υπάρχει σαφής αντίληψη πως η πολιτική είναι τα αφεντικά και βεβαίως έχουμε δύο ειδών ομάδες εδώ πέρα, τους κορυφαίους α, ε, α, ε, της διοίκησης και τους επιτρόπους που είναι ε, όλοι επαγγελματίες, αλλά σε τελική ανάλυση υπάρχει και η ξεκάθαρη αντίληψη πως η πολιτική είναι τα αφεντικά. Οπότε υπάρχει σαφής ιεραρχία. Αυτό σημαίνει βεβαίως πως έχουμε μία ομαλοποίηση θα έλεγα γίνεται πλέον φυσιολογική ε, ένα φυσιολογικό εκτελεστικό ε, σώμα θα λέγαμε ή ε, κομισιόν και ακριβώ η λογοδοσία αυτή κατέληξε σε μια διοίκηση η οποία μοιάζει όλο και περισσότερο με εθνική διοίκηση. Για να επανέλθω τώρα στο θέμα της οικονομικής λογοδοσίας, θέλω να πω πως αυτό το οποίο χρειαζόμαστε βεβαίως είναι ένα ζήτημα με περισσότερη ουσία αλλά και ε, περισσότερο βάρος ε, όσον αφορά την ε, λογοδοσία και έχει μειωθεί θα έλεγα λόγω της πολυπλοκότητας η διαφάνεια του συστήματος λογοδοσίας. Και βεβαίως το άλλο ζήτημα είναι το ότι έχουμε ένα, μια πολυεπίπεδη λογοδοσία, γιατί βεβαίως έχουμε και μια πολυεπίπεδη ε, διοίκηση, γιατί υπάρχει μια κοινή διαχείριση, ε, αλλά δεν μπορούμε να... Δεν μπορεί να λογοδοτήσει η Κομισιόν πέρα από το θεσμικό της ρόλο. Αλλά αυτό πρέπει να το δούμε. Καταλήγοντας. Είμαστε πάρα πολύ θετικοί θα έλεγα για το καθεστώς που υπάρχει όσον αφορά τη λογοδοσία. Οι θεσμικές αλλαγές ε, είναι αργές και δεν είναι κάτι το οποίο είναι μόνο θέμα διατάξεων. Βλέπουμε πως η διαδικασία αυτή συχνά είναι ζήτημα ερμηνείας ε, διατάξεων που πρέπει να ενεργοποιηθούν. Τα τελευταία δέκα χρόνια λοιπόν είχαμε αρκετά μεγάλη βελτίωση της λογοδοσίας εντός της ε, Κομισιόν. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mrs. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Βίλε. Ο Χουσέιν Κασίμ τώρα, από το Πανεπιστήμιο του East Anglia. Ναι, είναι βίντεο διάσκεψη. Ίσως ε, τα τεχνικά μέσα λειτουργήσουν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 Το δικό σας θέμα αφορά το ρόλο της, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σε σχέση με την προεδροποίηση ή συλλογικότητα. General. Um, essentially I've got four observations that I'd like to make. Um, the first is that the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 Thank you very much, Professor It's right away in the middle of the night. Uh, ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κασίμ. Ε, είναι ξημερώματα εκεί που βρίσκεστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ομιλία σας. Ε, η, η ποιότητα δεν ήταν η επιθυμητή. Δεν μπορούσαμε να ακούσουμε όλες τις λεπτομέρειες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καταλάβαμε την ουσία της παρέμβασής σας. Λοιπόν, Άρχεται η συζήτηση. Είναι καλύτερο να θέσουμε κατευθείαν ερωτήματα στον κύριο Κασίμια και τον έχουμε ακόμα μαζί μας. Κυρία Γκρέσλε. Thanks a lot for, uh, for, your, uh, for your speech and for the interesting results. Um,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 You can still follow the discussion. Perhaps if you want to make an intervention, we come back to you. But I now open the floor for the discussion and the questions to all the other panelists. Mr. Balchitis, you are very long on the list. Taip, ačiū, gerbiamas pirmininkė. Mes šiandieną tikrai turėjome progos daugelį dalykų išklausyti ir pirmiausia turbūt ε, yeah. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατάσταση, η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και σας ευχαριστώ για την πρωτοβουλία αυτή για μια για το να μιλήσουμε για μεταρρυθμίσεις που μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα. Ο κύριος Σεμπαστιανή μας είπε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα στον τομέα της ε, διοίκησης. Ε, και τη σχέση των γενικών διευθυντών με τη Γενική Διεύθυνση, η οποία δεν είναι δικό τους φέουδο. Και βεβαίως ε, τα συμπεράσματα που βγάλαμε είναι πως ε, δεν επαρκεί ο συντονισμός που υπάρχει τα μέσα δεν χρησιμοποιούνται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Προβλήματα πρέπει να δούμε. Η κυρία Βίλε πρέπει βεβαίως ε, να τονίσουμε πως ε, σήμερα μέρα βεβαίως ε, είναι λιγότερο πολιτικοποιημένη η υψηλόβαθμη της Κομισιόν, αλλά βεβαίως θα πρέπει να πούμε πως δεν μπορούν τόσο εύκολα να μεταρρυθμίσουν αυτούς τα θεσμικά όργανα. Και πρέπει να πούμε πως ναι, είναι και ζήτημα ισορροπίας και ελέγχου. Γι' αυτό πρέπει να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό πρέπει να θέσουμε τις βασικές αρχές της μεταρρύθμισης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων έτσι ώστε να προχωρήσει πιο γρήγορα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ πως πρέπει να τεθεί λοιπόν ένα πλαίσιο και να καθοριστούν οι βασικές αρχές που θα έπρεπε να στηρίξουμε βεβαίως. Και βεβαίως κάθε δύο χρόνια νομίζω πρέπει να κοιτάμε πώς πάει η μεταρρύθμιση αυτή. για να προχωρήσει βεβαίως. Σας ευχαριστώ. Um, I have a question. Ευχαριστώ. Ένα ερώτημα θα ήθελα να θέσω προς τον κύριο Μπέκερ ε, για την ε, πάρα πολύ ε, συνοπτική και καλή παρουσίασή σας. Είναι ο ρόλος βέβαια των μεσαίων στελεχών το θέμα μας. Είναι κάτι βέβαια το οποίο αναφέρετε κι εσείς στην παρουσίασή σας. Το λέτε και στη σύνοψη του εγγράφου σας, πώς θεωρείτε ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις επηρέασαν το βαθμό της γραφειοκρατίας και ειδικότερα την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υποθέτω ότι δεν θα είναι πολύ ωραία η απάντησή σας ε, σε αυτό το ερώτημα, αλλά θα ήθελα να ακούσω την ανάλυση και την ε, δική σας αξιολόγηση για τα δύο αυτά ερωτήματα. λίγο πιο λεπτομερώς. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ η κυρία Γκρέσλη και μετά ο Πιέρ Δύο ερωτήσεις έχω προς όλους. Θα ήθελα να ακούσω τι μας συμβουλεύετε, τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε για να ενισχύσουμε το σώμα των επιτρόπων. Γιατί κάποια πράγματα με ε, ανησυχούν. Έχουμε αυτό το οποίο δηλαδή μας είπε ο κύριος Μπέκερ, τον πίνακα 3 και τον πίνακα 4 και τον πίνακα 5 στην παρουσίασή του. Οπότε εμείς Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε με τη δουλειά μας. Από, αν δούμε πως ε, με όλον αυτό τον μηχανισμό τα δύο τρίτα των ηγετικών στελεχών θεωρούν πως όλοι αυτοί οι μηχανισμοί ελέγχου δεν έχουν κάνει τίποτα για τη δουλειά τους πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά το ζήτημα και να δούμε το τι, τι γίνεται. Δεν θέλουν να λένε και να δίνουν λογαριασμό για το τι κάνουν. Γιατί κρίνουν τόσο άσχημα αυτά τα μέσα που δημιουργήσαμε. Στον δε 5 πρέπει όλοι μαζί να δούμε το πρόβλημα που λέγεται συνεννόηση και διαβούλευση μεταξύ των υπηρεσιών. Και εδώ ευχαριστώ τον κύριο Σεμπαστιανή. Η διαβούλευση αυτή και στην ανώτερη και στη μέση διοίκηση είναι δύσκολη. Ναι, αυτό εδώ το, το πράσινο χρωματάκι. Έτσι, και εδώ πέρα δύο τρίτα πρακτικά μας λένε πως δεν ε, στέκει, δεν είναι δεν λειτουργεί καλά. Τι κάνουμε δηλαδή, πώς θα έχουμε συνοχή και τι μας συμβουλεύεται να κάνουμε. Ζων Πιεροντή, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ που οργανώσατε αυτή τη συζήτηση με την εισηγήτριά μας. Ευχαριστώ ε, τους προσκεκλημένους μας ε, που μας έκαναν τις παρουσιάσεις τους. Απλώς να σας πω για την ποιότητα της βιντεοδιάσκοψης. Εγώ νομίζω ότι σε έναν ε, ε, φορέα σαν το δικό μας, ακόμη και με περιορισμένες συζητήσει, ε, ακόμη και με βιντεοδιάσκεψη θα έπρεπε να είναι λίγο υψηλότερη ποιότητα, ώστε να μπορούν ε, και οι διερμηνείς μας να μας κάνουν τη διερμηνία παρά το γεγονός ότι δεν είναι παρόν ο ομιλητής. Τώρα, επί της ουσίας, οι υπάλληλοι τέθηκαν όχι εν αμφιβόλο, αλλά τέλος πάντων ήταν αντικείμενο συζήτησης. Εγώ πιστεύω ότι, κα, ότι αν, αν η διοίκηση ανέλαβε δράση, υπήρχε ένα πρόβλημα με, την, με το πολιτικό επίπεδο. Και πάντοτε το πολιτικό επίπεδο έχει μία εξουσία. Ε, στους ε, πολιτικούς οργανισμούς. Τώρα το θέμα δεν είναι κατά πόσο είναι ε, το Κοινοβούλιο ή οι κυβερνήσεις που έδωσαν το δικαίωμα αυτό στους υπαλλήλου. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι υπάρχουν κακές γνωμοδοτήσεις του ελεκτικού συνεδρίου εδώ και κάποια χρόνια, χωρίς να υπάρχει ψήφος, πρόταση για πρόταση μομφής στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το ε, συζητήσουμε νομίζω ε, εν ώψη των ευρωεκλογών. Μιλάμε για τη διαχείριση τα τελευταία 10 χρόνια, 2004 με 2014. Αλλά τα τελευταία 10 χρόνια υπήρξαν νέα, πολλά νέα στοιχεία ε, ε, ενιαίο νόμισμα, 13 νέα κράτη-μέλη, αποτυχία της ε, στρατηγικής της Λισαβόνας. Δεν μάθαμε τίποτε. Για ποιο λόγο τελικά αποτύχαμε. Ε, γιατί δεν υπάρχει καλή ε, συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, κρατών μελών. Επίσης, το δημοψήφισμα για τη συνταγματική συνθήκη το 2005 απέτυχε και το λέω, αν είχαμε κάνει το, το, τότε 25 δημοψηφίσματα, δεν θα είχε δημοψήφισμα αρνητικό μόνο η Γαλλία και η Ολλανδία, αλλά και άλλες χώρες. Δεν φταίνε λοιπόν μόνο οι Γάλλοι ε, η διάρθρωση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, πνέει τα λίστια για να το πω έτσι. Το θέμα της Τελωνιακής Ένωσης για παράδειγμα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε όμως εκθέσεις του Ελληνικού συνεδρίου που μας λένε ότι δεν δουλεύει καλά γιατί οι εθνικές διοικήσεις ασκούν την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θέλουμε λοιπόν να έχουμε ε, μια τελωνιακή ένωση, γιατί δεν έχουμε μια τελωνιακή ένωση ε, που να ε, είναι υπεύθυνη Ευρωπαίοι υπάλληλοι, υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υπάλληλοι που θα δρούν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφορετικά πάντα θα υπάρχει χάος και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να προχωρήσουμε. Για το θέμα τώρα της κοινή διαχείρισης, εμένα θέλω να μου πούν την άποψή τους και οι πολιτικές ομάδες αλλά και οι προσκεκλημένοι μας. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Εξακολουθούμε να κάνουμε κατανομή ανακράτος μέλος. Κάθε κράτος μέλος ε, ε, ε, ακολουθεί το I want my money back των Βρετανών ε, και είδαμε ότι ήταν αδύνατο για μια κυβέρνηση να ε, ε, να σταθεί στο ύψος του ευρωπαϊκού του καθήκοντος ε, για να επιστραφούν ακριβώς αυτά τα λεφτά. Εγώ τι να σας πω, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, οικονομική της διαχείριση, εφόσον έχουμε εκτελεστικές υπηρεσίες για την οικονομική διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε προς μια Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να πλήξουμε την κυριαρχία των κρατών μελών. Δεν είναι η χρονική στιγμή να πειράξουμε μια ισορροπία που ήταν δύσκολο να την επιτύχουμε μεταξύ ε, των ε, εθνικών και των ευρωπαϊκών αρμοδιοτήτων, αλλά τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, έχει πλήρη τις αρμοδιότητές της, να τις ασκεί στο πλαίσιο ενός δημοσίου αξιώματος, αφήνοντας στα κράτη-μέλη τη φροντίδα της διαχείρισης των εθνικών τους ευθυνών και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταλάβει ότι τουλάχιστον ε, τα τελευταία 6 με 10 χρόνια ε, είναι ας πούμε μια θηγατρική ε, των κρατών μιλών και όχι το αντίστροφο. Όπως είπατε και εσείς κυρία Βίλε, πρέπει να αποεθνικοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω εσείς κυρία Βίλε το είπατε, αλλά πρέπει να δούμε τι λένε και οι πολίτες. Στη συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπεται αυτή η αποεθνικοποίηση, γιατί θα έπρεπε να μειωθεί ο αριθμός των επιτρόπων. Όμως η Δηλαδή μας είπαν ότι αν εγώ, αν εμείς δεν έχουμε ε, ε, δεν έχουμε επίτροπο, ε, δεν θα δεχθούμε να τεθεί και πάλι σε δημοψήφισμα η συνθήκη της Λισαβόνας. Οπότε επανήλθαμε στο ένα επίτροπο σαν κράτος μέλος. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να συμφιλιώσουμε κάποτε τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συγγνώμη που μακρηγορώ. Για να επανέλθω λοιπόν στον έλεγχο και την εκτέλεση του προπολογισμού, προτείνω να κάνουμε τουλάχιστον μία μελέτη για την κατάργηση της κοινή διαχείριση. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλος τον λόγο. Θα ήθελα κι εγώ να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα ακούσαμε πως εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα προηγούμενα χρόνια υπάρχει μια ευρωπαϊκή κουλτούρα που αναπτύχθηκε είτε σκεμμένα είτε εκ των πραγμάτων Και βέβαια ακούσαμε το τι γίνεται και με το προσωπικό από τις νέες χώρες όπου καθένας βεβαίως ε, κουβαλάει μαζί του τη δική του διοικητική ε, κουλτούρα. Οπότε τίθεται και εδώ το ερώτημα του τι ε, αντίληψη έχουμε για την διοίκηση. Υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις. Εάν δείτε παραδείγματο χάρη τη χώρα μου, την ε, Γερμανία, υπάρχει μία διοίκηση ε, εξειδικευμένη, η οποία ιδεοδός ε, δρά ανεξάρτητα από την πολιτική και κατευθύνεται από τους πολιτικούς ε, προϊσταμένους, οι οποίοι αλλάζουν με τις εκλογές. Αν δούμε το αμερικανικό μοντέλο, και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες που ακολουθούν κάτι άλλο. Εκεί πέρα μεγάλα τμήματα της διοίκησης αλλάζουν όταν αλλάζει η κυβέρνηση. Οπότε μπορούμε να πούμε πως υπάρχει μια πολιτική κατεύθυνση της διοίκησης. Οπότε η υπόθεση αυτή πως έχουμε μια ανεξάρτητη διοίκηση η οποία θα δρά απολυτικά δεν στέκει. Τώρα εγώ δεν θέλω να αξιολογήσω ποιο είναι το καλύτερο. Ακούσαμε τους δύο επιτρόπους ε, και πως ε, καμιά φορά είναι δύσκολη η πολιτική κατεύθυνση όταν αναπτύσσεται μια εσωτερική ζωή στη γραφειοκρατία και δεν αναγνωρίζει καμιά φορά η γραφειοκρατία πως οι αποφάσεις έχουν πολιτική διάσταση. Και βέβαια το ακριβώς αντίθετο θέλουμε, γιατί δεν είναι πολιτικά επιθυμητό ή και από τους πολίτες ε, έτσι, διορισμένοι γραφειοκράτες, για να το πω υπερβολικά, να λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις και να μην το κάνουν αυτό οι αιρετοί. Οι αιρετοί που δίνουν και λόγο, έτσι, οι πολιτικοί. Και αυτό βεβαίω είναι ένα τμήμα του δημοκρατικού ελέγχου, γιατί υπάρχει βεβαίω και η λογοδοσία των πολιτικών. Επέναντι στους πολίτες, το λαό, στη θεωρία τουλάχιστον. Και εδώ πέρα είναι το ερώτημά μου. Και εδώ είναι το ζήτημα προς τον κύριο Μπέκερ. Μιλήσατε για το θέμα της αποκέντρωσης. Έχουμε, όπως είπαμε, αυτή την αποκεντρωμένη ευθύνη για τους φόρους, την οποία συζητήσαμε σε διάφορα επίπεδα και εδώ πέρα εφαρμόζεται βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εσείς επίσης διαπιστώνετε πως απαιτείται κάποιος συντονισμός. Ίσως λοιπόν θα μπορούσατε κι εσείς από τη δικιά σας σκοπιά να μας πείτε αν σας κατάλαβα καλά, λέτε πως δεν αμφισβητείτε επί της αρχής η αποκέντρωση, αλλά ζητάτε καλύτερο συντονισμό. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες συμβουλές το, ή να μας πείτε σε ποια κατεύθυνση πάει. Δηλαδή είναι, ε, βασίζεται σε αποτελέσματα, σε επιδόσεις, ε, αυτά που μας είχαν αποσχολήσει στο παρελθόν. Εμείς θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια σχετικά πράγματα. Τα ερωτήματα νομίζω απευθύνονται σε όλους τους παρόντες. Προτείνω να ξεκινήσουμε με τη σειρά των ομιλητών. Οπότε να δώσω το λόγο στον κύριο Μπέκερ πρώτα και μετά τον κύριο Σεβαστιανή, την κυρία Βίλη και τον κύριο Κασίμ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γερμανικά. Το πρώτο ερώτημα, αν κατάλαβα καλά, ήταν αφορούσε την ισορροπία της γραφειοκρατικοποίησης και της αποτελεσματικότητας μεταρρύθμισης. Τι εννοούμε όμως εδώ πέρα, γιατί η γραφειοκρατικοποίηση σημαίνει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα μέσω των ε, διαχειριστικών σχεδίων παραδείγματος χάρη. Μετά λέτε ναι, πως η δουλειά κάποιον έχει γίνει αποτελεσματικότερη. Από την άλλη όμως μπορούμε να έχουμε και υπερβολικά πολλές τυπικές απαιτήσει. Ανέφερα το παράδειγμα των τμήματαρχών. Πράγματι, θα πρέπει και η πολιτική του προσωπικού να βασίζεται στις επιδόσεις και όχι μόνο στην αρχαιότητα. Και μετράνε βεβαίως οι τμήματάρχες τις ε, επιδόσεις. Αλλά μετά μας λένε παιδιά δεν, κάνω τίποτα άλλο, όλο με το προσωπικό ασχολούμαι. Ε, δηλαδή πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Τα είχαμε παραμελήσει λίγο και ίσως τώρα υπερδιορθώσαμε προς την άλλη κατεύθυνση. Και βεβαίω πρέπει να πω πως πρέπει πράγματι να ξέρουμε πού βρίσκεται ο καθένας, σε τι δουλειά κάνει και το άλλο ζήτημα είναι πως πρέπει να πούμε πως πρέπει να έχουμε μια πάρα πολύ ε, προσεκτική τοποθέτηση στο ζήτημα αυτού του συντονισμού γιατί όπως σας είπα συχνά οι μεταρρυθμίσεις ε, δεν είναι και τόσο δημοφιλείς στους ανθρώπους που τελικά πρέπει να τις εφαρμόσουν και πρέπει να είμαστε κάπως λίγο προσεκτικοί αυτό ως προς αυτή την ερώτηση τι άλλο. Για τα μέσα τα ίδια το είπε η κυρία Γκρέσλε. Αν δείτε το τι γίνεται και το εάν διευκολύνεται η καθημερινή εργασία με τον τρόπο αυτό. Εντάξει, βλέπετε πως τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά, έχουν απαντήσει διαφορετικά οι άνθρωποι, αλλά αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι πως οι υποχρεώσεις αυτές ε, αναφοράς, συνεχούς αναφοράς, θεωρούνται κάτι το οποίο κάνουν οπωσδήποτε ε, οι άνθρωποι, αλλά δεν το θεωρούν μέρος της δουλειάς τους, δεν ότι αυτή είναι η δουλειά τους. Και Επίσης ο βαθμός λεπτομέρειας των αναφορών αυτών είναι σημείο κριτικής. Αλλά όπως είπα το σχέδιο αυτό το διαχειριστικό σχετικά θετικά το βλέπουν οι γενικοί διευθυντές ε, και εκεί πέρα μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε το τι, το τι θέλουμε και μπορούν και αυτοί βεβαίως να το μεταδώσουν μετά στους υφισταμένους τους. Οπότε... Ναι, είναι και το ζήτημα πράγματι του πώς ε, συμβιβάζονται οι στόχοι της κάθε γενικής διεύθυνσης με τη γενική εικόνα. Σας ευχαριστώ κύριο Σεμπαστιανή. Δεν ξέρω αν χρειάζεται. Επιβεβαιώνω πάντως ε, απόλυτη την ανάλυση που έγινε για την αντίληψη και το ρόλο του τμήματάρχη με, πριν και μετά την μεταρρύθμιση είναι χάνη στην κατανομή ευθυνών. Είναι μια επιλογή που έγινε να κοπεί ο δεσμός μεταξύ του συντονιστικού ρόλου της ομάδας και των τεχνικών ικανοτήτων που πρέπει να έχει κάποιος για να είναι αξιόπιστος όλο το πλαίσιο διαχειρίστηκε, περιορίστηκε στη διαχείριση πόρων. Δεν είναι ασήμαντο μένα, αλλά βρισκόμαστε τώρα σε ένα πλαίσιο όπου ο τμηματάρχης περνάει το χρόνο του κάνοντας αυτό που περιγράφεται, χωρίς να μπορεί όμως να καταλάβει την τεχνική εμβέλεια των φακέλων που πρέπει να διαχειριστεί. Και αυτό δημιουργεί ε, τεράστια απώλεια γνώσης και ε, εμπειριών. Κάθε πρέπει να αρχίσει να, με, να μελετάει όλες τις ε, δραστηριότητες, όλη την ομοθεσία για άδειες, άδειες αναποδοχών, για να μπορέσει να εφαρμόσει με συνεκτικό τρόπο το κείμενο και να μην έχει ερμηνεία δική του. Πρόκειται για πραγματικά σημαντική απώλεια ικανοτήτων που μας λείπει. Καλό θα ήταν να κλείσει. Για το δεύτερο θέμα, τη σταδιοδρομία του υπαλλήλου που συνδέεται με προσωπικές ή πολιτικές σχέσεις. Όλοι έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχει ένα είδος spoil system, κρυμμένο spoil system, που καταγγέλουμε και ορίζουμε ως αλεξιπτωτιστές. Αυτό αποσταθεροποιεί τη λειτουργία των υπηρεσιών και επιπλέον δημιουργεί το, την εντύπωση ότι για να προχωρήσεις πρέπει να σε εκτιμήσει ένα άτομο. Όχι αναγκαστικά να σε εκτιμήσουν γιατί μπορείς να δουλέψεις καλά. Τρίτον, για την ε, ενδοϊπηρεσιακή διαβούλευση. Νομίζω ότι αυτό που γίνεται για την υλοποίηση της αποκέντρωσης των ερευνητικών προγραμμάτων είναι ένα τέλειο παράδειγμα οι τρει κεντρικέ υπηρεσίες, όχι οι γενικοί διευθυντέ που έχουν την ευθύνη τη εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων, οι τρει κεντρικέ υπηρεσίε, η Γενική Γραμματεία, η Γενική, Γραμματεία, Γενική Διεύθυνση Διοίκηση και η Γενική Διεύθυνση προπολογισμού, οργανώνουν μία διυπηρεσιακή διαβούλευση με την πολιτική επιταγή των δύο πολιτικών Σεύκοβιτς Λεβαντόφσκι για να ετοιμάσουν μια ανακοίνωση καπέλο πλαίσιο που δίνει το ευρύ πλαίσιο στην, ε, στην Επιτροπή για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Στο κείμενο αυτό προβλέπουμε πέντε κεντρικές υπηρεσίες για τη διαχείριση των προγραμμάτων και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία. Η λογική αυτή πρέπει να εφαρμοστεί, διότι ενισχύει το αίσθημα κάθε υπαλλήλου να μετέχει σε έναν οργανισμό που μπορεί να συντονίσει και να διαχειριστεί τις διαφορές. Αυτό που λείπει είναι η ικανότητα να βρεθεί η δυνατότητα επίλυσης των διαφορών μεταξύ γενικών διευθύνσεων για παράδειγμα και αυτό μπορεί να γίνει από υπηρεσίες κεντρικού επίπεδου που έχουν συγκεντρωτική εικόνα και προσβλέπουν στο συμφέρον της υπηρεσίας και όχι των κλάδων ή των μεν και των δε. Τέτοιες οργανώσεις θα μας επιτρέψουν να έχουμε αξιόπιστους συνομιλητές που σίγουρα θα μπορούν να βελτιώσουν τα καταστροφικά αποτελέσματα του 70 και θα επιτρέπει ο υπάλληλο να μην αισθάνεται ότι είναι ιδιοκτησία του κάθε προϊσταμένου του. Αυτό είναι ο σωστός δρόμος και πιστεύω ότι η δική σας συμβολή είναι σημαντική στις αλλαγές αυτές. Ευχαριστώ. Κύριε κυρία αν έχετε ερωτήσεις. κυρία Βίλε, αν έχετε, πιστεύετε ότι μπορείτε να απαντήσετε, ότι θέλετε να απαντήσετε. Για τη συλλογικότητα. Άλλο θέμα είναι η συλλογικότητα. Σε μια επιτροπή 28 επιτρόπων και όχι 6. Αυτό είναι αναπόφευκτο, δηλαδή θα υπάρξει μια προεδροποίηση, συγκεντρωτική προσέγγιση. Η συλλογικότητα προφανώς εξυγχρονίστηκε γιατί έχουμε και το πολιτικό πλαίσιο της πενταετής καθοδητήριας γραμμές που είναι σημαντικές για την Επιτροπή μπορεί να τα παρουσιάσει στο τέλος του, των πέντε ετών. Άρα ο πρόεδρος έγινε πιο, απέκτησε μεγαλύτερη δυνατότητα επιρροής. Ε, Και μην ξεχνάτε ότι η συλλογικότητα ε, σχετίζεται με το workflow Μιλάμε για το διοικητικό επίπεδο, το managerial, αλλά όχι το επίπεδο των ιδιαίτερων γραφείων των επιτρόπων, όπου γίνεται πολύ, διαμορφώνεται σημαντική πολιτική και εκεί διαμορφώνεται και το πνεύμα της ε, συλλογικότητας. Εγώ θα πρότεινα, το, θα έλεγα μάλλον, ότι το επίπεδο των προσωπικών γραφείων μπορεί να βελτιωθεί και να αποκτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια. Κάτι άλλο η απεθνικοποίηση. Οι εδαφικές αρχές ε, ή ο αλεξιπτωτισμός μειώθηκε. Εμείς λέμε ότι τα ιδιαίτερα γραφεία και το ανώτερο επίπεδο της διοίκησης έγιναν πολύ πιο πολυεθνικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε τελείως σε απεθνικοποίηση. Οι εθνικές τομές είναι σημαντικές στην ευρωπαϊκή πολιτική. Κάθε κράτος μέλος θέλει να έχει εκπροσώπηση στην Επιτροπή. Λογικό είναι. Διότι μιλάμε για ένα πολιτικό εκτελεστικό όργανο. Δεν θα έλεγα λοιπόν ότι η εθνικότητα δεν παίζει ρόλο. Αλλά υπάρχουν διαδικασίες απεθνικοποίησης στη διοίκηση, σε επίπεδο προσωπικών γραφείων που οδήγησαν σε πιο πολυεθνική οργάνωση. Η γαλλογερμανική κουλτούρα, η παλιά γαλλογερμανική κουλτούρα με τις διάφορες διευρύνσεις προς Αγγλία, προς Σκανδιναβία άλλαξε δημιουργήθηκε μια διοικητική κουλτούρα, νέες δομές λογοδοσίας και έκαναν την Επιτροπή το πιο πολυεθνικό όργανο στην Ένωση. Τέλος, θα έλεγα ότι οι ρυθμίσεις λογοδοσίας εστιάστηκαν και από την Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο μόνο στον έλεγχο της Επιτροπής. Υπάρχει και η λογοδοσία προς τον ψηφοφόρο, έξω από εδώ. Έχουμε εκλογές το Μάιο, που θα είναι 28 εκλογές, όχι μία πανευρωπαϊκή εκλογή. Αυτό είναι κρίμα, διότι οι εκλογέ είναι εκλογέ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά δεν φαίνεται ότι η σύνθεση της Επιτροπής θα αντικατοπτρίζει την σύνθεση του Κοινοβουλίου. Άρα και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα λογοδοσίας που πρέπει να προσέξουμε. Ευχαριστούμε.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 Πλην δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, ο κύριος Σεύκοβιτς, αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έμεινε μαζί μας, μας τιμά ιδιαίτερα αυτό, κάτι το οποίο δείχνει ενδιαφέρον ε, για αυτά που συζητούμε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, το εκτιμούμε ιδιαίτερος και θα ήθελα να σας δώσω τη δυνατότητα να σχολιάσετε ορισμένα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ ε, για τα καλά σας λόγια και εγώ θα ήθελα να συνοψίσω λέγοντα να ευχαριστώ πάρα πολύ τους καθηγητές, ακαδημαϊκούς, ε, ε, ερευνητές και αναλυτές για όλα τα θετικά σχόλια που έκαναν ε, για τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια. Δεν άκουσα μόνο εσάς, γιατί ξέρω ότι υπήρξαν και άλλες ε, προτάσεις ε, για το πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα και δεν αφορούσαν αυτά μόνο εμένα, αλλά ε, και τα μέλη της Επιτροπής σας που άκουσαν πολύ προσεκτικά τις προτάσεις και τα σχόλιά σας. Θα δουλέψουμε πολύ σκληρά να δούμε πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε σε καθημερινή βάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και εσάς και την κυρία Γκρέσλε για την οργάνωση αυτής ακρόασης, γιατί μας επιτρέπει να ε, μαθαίνουμε περισσότερα, να ε, ξέρουμε τι μας γίνεται, να βελτιωνόμαστε και θα εξασφαλίσω ότι θα μεταφερθεί το μήνυμα ότι τα χρήματα δαπανώνται σωστά, ότι είναι προσανατολισμένα περισσότερο προς τις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών και ότι η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιάνει τόπο και για τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους πολίτες της. Θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια σε σχέση με την ερώτημα για τη συλλογικότητα, πώς μπορεί κανείς να την ορίσει. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις παρεμβάσεις. Να σας πω ποια είναι η δική μου πρόταση. Καταρχά, ε, εκτιμώ όλο ιδιαίτερω την παρέμβαση που είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Επίτροποι πρέπει να ενδιαφέρονται για την δουλειά των συναδέλφων του. Δεν είναι κανεί υπεύθυνο μόνο για το δικό του χαρτοφυλάκιο και για τα δικά του θέματα. Συχνά ε, όταν ε, είναι λίγο διαφορετικό το ε, ιστορικό του καθενός, η διαχείριση που κάνει είναι λίγο διαφορετική. όταν είναι δύσκολη καιρή είναι πάρα πολύ σημαντική η αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ των επιτρόπων ε, και η παρουσίαση κοινών γραμμών που μερικές φορές καθίστανται ιδιαίτερα δύσκολη όταν πρέπει κανείς να εξηγήσει ε, κανείς μια δύσκολη πολιτική που έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό στη χώρα του ε, και πρέπει να το κάνει με καλή πιστή γιατί μερικές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο να λάβει κανείς τη σωστή απόφαση για δύσκολα θέματα. Η συλλογικότητα βέβαια δεν εξαντλείται εκεί που ε, συνεδριάζει το Σώμα των Επιτρόπων. Είναι μια πραγματικά ευρύτερη δουλειά ε, με την καθοδήγηση των γενικών διευθυντών που μας βοηθούν πάρα πολύ και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι πραγματικά να συντονίζουν τη δουλειά τους μαζί μας ώστε το αποτέλεσμα ε, μετά που βγαίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι ένα αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Όσον αφορά τώρα τα θέματα των μεσαίων στελεχών τα οποία αναφέρατε, είναι γεγονός ότι οι τμηματάρχες είναι εξαιρετικά απασχολημένοι άνθρωποι. Γιατί, γιατί 16 υπαλλήλου έχουν ε, ω υφισταμένου ε, και πρέπει να γίνουν προσωπικές συζητήσει, πρέπει να γίνουν αιτήσει εκθέσεις, πρέπει επίσης... Ε, να ε, ληφθεί υπόψη και η σταδιοδρομία των ε, ε, υπαλλήλων σου γιατί δεν είσαι μόνο υπεύθυνο για το τι βγαίνει από το τμήμα σου αλλά είσαι υπεύθυνο και για τους υφιστάμενούς σου. Οπότε αυτό σημαίνει βέβαια πολύ χαρτούρα. Δεν είναι πάντοτε πάρα πολύ εύκολο να διεκπαιρεώσει κάποιο όλα αυτά τα καθήκοντα, αλλά προσπαθούμε να απλοποιήσουμε ορισμένα πράγματα όσον αφορά την ετήσια αξιολόγηση, για παράδειγμα. Θα δούμε πώς ε, θα το κάνουμε στο μέλλον. Ε, υπάρχει μια διαφορετική νοοτροπία. Το σύστημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι λίγο διαφορετικό από το σύστημα του Κοινοβουλίου του Συμβουλίου. Αυτό το οποίο επίσης ε, συγκρατώ από τα σχόλιά σας είναι ότι μερικές φορές τα μεσαία ε, διοικητικά στελέχη είναι οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν αυτή τη θέση γιατί θεωρούν ότι αυτή είναι μια πρόοδος στην καριέρα τους, ότι πρέπει να πάρουν αυτή τη διοικητική θέση αν θέλουν να προχωρήσουν στην ε, καριέρα τους είναι κάτι για το οποίο πρέπει να έχουμε νομίζω περισσότερες επαφές μαζί σας για να εξευρεθεί μια σωστή ισορροπία. Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε αυτούς τους συμβουλευτικούς ρόλους, γιατί πολύ συχνά χρειαζόμαστε τους εμπειρογνώμονες μας, εξαιρετικούς νομικούς, εξαιρετικούς οικονομολόγους, εξαιρετικούς ειδικού στον τομέα τους που θέλουν να ε, προχωρήσουν ε, στην εμπειρογνωμοσύνη τους όμως, στον τομέα της εμπειρογνωμοσύνης τους ε, και θεωρούν ότι δεν θα ήταν πάρα πολύ καλή διοικητική. Πρέπει λοιπόν να έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν αυτή τη δυνατότητα εξέλιξης προσωπικής τους καριέρας στη δική τους εμπειρογνωμοσύνη και να μπορούν να μας δίνουν καλές συμβουλές, να δίνουν καλές συμβουλές στους ανώτερους διοικητικούς. Όσον αφορά τώρα τον συντονιστικό ρόλο των προέδρων. Να σας πω από την πείρα μου οι επαφές μεταξύ των ε, επιτρόπων είναι συχνές. Αν εγώ δω ας πούμε ότι έχω ένα σοβαρό πρόβλημα ε, γιατί κάποιος γενικός διευθυντής δεν μπόρεσε να φτάσει σε συμφωνία και πιστεύω ήδη καταλαβαίνω από τις διπηρησιακές ε, συζητήσεις ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα, προσπαθούμε πράγματι να συζητήσουμε πολύ και να βρούμε μία λύση. Είναι σπάνιο να είναι έντονες οι διαφορές στις συζητήσεις του Σώματος των Επιτρόπων, γιατί συζητούμε μεταξύ μας τακτικά, οι ομάδες μας είναι σε συνεργασία και έτσι ξέρω ότι, και ξέρω και εγώ ότι είμαι σε μια πολύ καλή ε, ε, συναδελφική σχέση με τους υπολείπους επιτρόπους. Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούμε να αποφασίσουμε ε, με συνένεση και να υπερασπιστούμε την κοινή γραμμή του Σώματος των Επιτρόπων. Τελευταίο σχόλιο, γιατί επίσης ε, αναφέρεται συχνά αυτό το θέμα... Ε, τον αλεξιπτοτισμό Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προσπάθησε να σας το εξηγήσω και αυτό στις, ε, στα ενακτήρια μου σχόλια. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα τελευταία 10-15 χρόνια λόγω των νέων ευθυνών, ε, λόγω της διεύρυνσης, αλλά παράλληλα ε, πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα πρόσληψης κάποιου εξωτερικού, αν χρειάζεται η εμπειρογνωμοσύνη. Ε, για παράδειγμα, οι προσωρινοί κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, έχουν ε, ε, πάρα πολλές δυνατότητες να γίνουν ε, ε, υπάλληλοι της Ένωσης βάσει της πρώτης αξιολόγησής τους, βάσει διαγωνισμών. Προσπαθούμε να θέσουμε κάποια κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν ώστε να εμπλουτίσουμε τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σημαντικό να έχουμε τα απαραίτητα ταλέντα να, ε, να προχωρήσουμε. Όσον αφορά τις ομάδες, ε, έχει δίκιο η κυρία ε, Βίλε κάθε ομάδα, αν μιλάω για τα μέλη της ομάδας του κάθε επιτρόπου που εκπροσωπούν ε, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, τους ε, επιτρόπους, υπάρχει μια σαφής γραμμή που ακολουθείται, τουλάχιστον τρεις εθνικότητες πρέπει να εκπροσωπούνται και η μισή πρέπει να είναι υπάλληλοι. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια συνέχεια ότι υπάρχει συνοχή και όπως είπατε και στην πράξη λειτουργεί καλά το σύστημα αυτό. Είμαστε πολύ Ευρωπαίοι στο, ως προς τη σύνθεση των ομάδων μας. Να σας ευχαριστήσω μία ακόμη φορά κύριε Πρόεδρε για την πρόσκλησή σας. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή σας που ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ε, έχει καλύτερες επιδόσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ελπίζω του χρόνου να φανεί αυτό όταν θα πρέπει να ψηφίσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ε, να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους προσκεκλημένους μας που μας έδωσαν πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες για το πώς μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σεύκοβιτς. Όχι μόνο εκτιμούμε την παρουσία σας εδώ, αλλά Εκτιμούμε και την ανακοίνωση ότι θα λάβετε υπόψη αυτά τα οποία εμείς ως Επιτροπή ε, σας δίνουμε ως πληροφορίες, όπως επίσης και οι ε, επιστήμονες που ήταν εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ για να ολοκληρώσουμε την ακρόασή μας. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπανε. Έμαθα μια νέα λέξη, upstream coordination. Θα προσπαθήσω να μάθω και τι σημαίνει. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Άνταμσεν επίσης της γραμματείας με τον οποίο ε, οργανώσαμε την ακρόαση αυτή. Και αυτοί που δεν ήθελαν να λάβει χώρα θέλουν να μου πούν γιατί. Γιατί νομίζω πως τα σημερινά αποτελέσματα ήταν θετικά. Με σημαντικά ευρήματα. Δεν ξέρω, ίσως όλα αυτά να είναι μία όψη του νομίσματος και να προσπαθεί η διοίκηση να υπερβεί ζητήματα που προέκυψαν με την αποκέντρωση κτλ. Και βεβαίως ε, να δούμε πως ε, η διοίκηση εφαρμόσει με συνοχή την πολιτική. Βεβαίως το θέμα με εμένα είναι και τα μέσα που έχουν αποδειχθεί ότι δεν λειτουργούν. Είναι παλαιό το πρόβλημα. Καλό νομίζω λοιπόν κάποιες διαδικασίες να τις επανεξετάσουμε. Να δούμε και το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας Κομισιόν. Τώρα η αξιολόγηση του προσωπικού είναι εσωτερικό ζήτημα της Κομισιόν. θα πρέπει νομίζω να προσπαθήσουμε να δούμε τι γίνεται και εκεί πέρα. Τώρα για το πώς θα εμπλακούν οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες στη διοικητική αυτή ε, ζωή. Γιατί τα πολλά περιστατικά που είχαμε νομίζω με οδηγούν στο ότι πρέπει να ενταχθούν στις διαδικασίες της Κομισιόν. Επίσης, ένα ζήτημα δεν ακούστηκε το τι θα πρέπει να κάνουμε από εδώ και μπρος τη γραμμή πρέπει να ακολουθήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή τη συλλογικότητα της Κομισιόν και από πλευρά συντρόφων. Αυτά. Και σας ευχαριστώ όλους και νομίζω όλα αυτά θα τα αναφέρω και σε ένα έγγραφο εργασίας. Σας ευχαριστώ κυρία Γκρέσλε. Ήθελε η Επιτροπή μας να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Οι φόβοι βεβαίως αποδείχθηκαν μη δικαιολογημένοι. Ευχαριστώ και εγώ τα μέλη του πάνελ, τους κυρίους Μπέκερ, Κασίμ ε, και λοιπούς και τον ε, κύριο Σεύκοβιτς. Σας ευχαριστώ για το ότι μείνατε και για τις παρατηρήσεις σας. Άρα τελειώνει η ακροασή μας, διακόπτεται η συνεδρίαση. Θα συνεχίσουμε στις 3 ώρα το απόγευμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Καλό το απόγευμα.